Please, um, apologies for that. Please, can we adopt the agenda? Παρακαλώ, καθίστε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσει τη Πρόεδρου. Να σας πω ότι η έκθεση για την αποστολή στην Ολλανδία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Στο σημείωμα προ τα μέλη και διατίθεται και στην ιστοσελίδα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στην ιστοσελίδα. Πολύ ωραία. Μεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίασή μα και αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ε, εφαρμογη ή e-meeting για να τα παρακολουθήσετε ε, και από τον υπολογιστή σας ή από την ταμπλέτα σας. Έχετε και μια νέα έκδοση του newsletter και εξακολουθώ να λαμβάνω πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ενστάσεις για τα πρακτικά. Αν δεν διατυπωθούν λοιπόν ε, αντιρρήσει μέχρι τέλη τη συνεδρίαση την Πέμπτη, θα, θεωρούμε, θα θεωρήσουμε την εγκεκριμένα. Θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για τι δύο τριμερεί διαλόγου που διεξαγάγονται από τον Ανδρέα Σουάπ και οι δύο παρακολουθούνται για την ασφάλεια πληροφοριών και για τις ιατρικές συσκευέ. Θα θέλετε να μας ενημερώσετε για το πώς έχει κατάσταση και για τις δύο αυτούς τριμερείς διαλόγου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια, αλλά αυτό το κοπλιμέντο θα έπρεπε πραγματικά να το μεταβιβάσω στους υπαλλήλου και της ομάδας και της Επιτροπής. Γιατί διαπραγματευόμαστε με την Λουξεμβουργιανή Προεδρία και είναι η τρίτη Προεδρία στο καινούριο κοινοβούλιο, στην καινούργια θητεία και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκαθαρίσαμε με σαφήνεια το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε και πολλά τα παρακολουθούμε με επιμονή και υπομονή και θα μπορέσουμε να τα επιβάλλουμε. Θα υπάρξουν λοιπόν δύο τομείς ένα παράρτημα δύο, έτσι διαμορφώνεται η διαπραγματευτική μας θέση για τις υπηρεσίες της οικονομίας offline δεδομένα τα οποία αφορούν ψηφιακά στοιχεία της διαδικασίας και θα διαμορφωθούν από τους παρόχους για να είναι ανθεκτικά, να είναι δηλαδή ασφαλή από κυβερνοεπιθέσεις και στο νέο προσάρτημα 2α θα υπάρχει ένα μικρό τμήμα των ψηφιακών παρόχων υπηρεσιών στον τομέα εφαρμογής, όχι επειδή αποτελούν κρίσιμες υποδομές, αλλά επειδή αφορούν τις κρίσιμες υποδομές των ψηφιακών στοιχείων, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και αυτά να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας. Τρεις τομείς λοιπόν θα υπάρξουν, τρεις ε, ψηφιακοί πάροχοι ε, τρεις κατηγορίες ψηφιακών παρόχων, οι οποίοι τα ληφθούν υπόψη. Καταρχάς έχουμε τις online πλατφόρμες ε, αγοράς, ε, ένα τομέα το οποίο το κοιτάξαμε και στην κανονισμό για την επίλυση διανέξεων της κυρίας Τόν. Και εδώ θα καλύπτονται πολλά είδη ψηφιακών πλατφόρμων, αλλά όχι τα C2C όπως ονομάζονται. Θα υπάρχουν και ένας δεύτερος τομέας, ε, οι μήχανες αναζήτησης, όπου θα ξεκαθαρίσουμε με νομικό τρόπο τι ε, ψηφιακές, τις ε, μηχανές αναζήτησης μπορούν να χρησιμοποιούν τα κανάλια αυτά, προκειμένου να είναι και να παραμείνουν σίγουρες και ο τρίτος τομέας, ο οποίος είναι στον τομέα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ήτρε, όπου και πάλι έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Ντέλκα στη Γιοβέρα, θα ασχοληθεί με το θέμα του νέφους, του cloud. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την οδηγία και ο στόχος της οδηγίας είναι οι πάροχοι, οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών να είναι υπεύθυνοι για θέματα ανθεκτικότητας, προστασίας δηλαδή, και όταν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο κίνδυνο, όταν εντοπίζουν κάποιο κίνδυνο, να το κοινοποιούν στις εθνικές αρχές με απότερο σκοπό να υπάρχει συντονισμένη κοινή δράση πρόληψης και καταστολής εφόσον αυτή κρυφτεί απαραίτητη. Τα τελευταία λοιπόν στοιχεία θα πρέπει να τα συζητήσουμε με το Συμβούλιο κυρία Πρόεδρε για το κατά πόσο θα καταφέρουμε στις ψηφιακές ε, υπηρεσίες να πετύχουμε μια πλήρως εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση αλλά από ό,τι φαίνεται τα μέλη ε, έχουν την προθυμία αυτή. Γιατί φαίνεται να το κάνουν αυτό. Γιατί καταλαβαίνουν ότι μόνο εφόσον υπάρξει κανονιστική ομοιομορφία θα μπορέσει να υπάρχει ευρωπαϊκή προσέγγιση και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε να μην περιοριστούμε στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή αλλά να βρούμε κάτι το οποίο να βγάζει νόημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την ε, βοήθεια τη δική σας και τη βοήθεια των ε, σκιωδών, δεν είναι εδώ πέρα ούτε ο κ. Γκρουντ και ο κ. Άλμπρεχτ από τους πράσινους, Είμαστε όμως σε καλό δρόμο και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό σας έδωσα μια καλή επισκόπηση του που βρισκόμαστε στην παρούσα φάση. So Συνοψίζοντας λοιπόν, σας ευχαριστούμε Ανδρέας. Ο επόμενος διάλογο, διάλογος έχει πραγματιστεί για σήμερα το βράδυ. Και εγώ θα ενημερώσω την Επιτροπή την Πέμπτη. Δυστυχώς δεν θα είστε εδώ, αλλά θα μεταφέρω τα όσα λιμήφθησαν εκεί. Ήταν εξαιρετικά ενδελεχής η εξέταση και η διαπραγμάτευση για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο ή να προχωρήσουμε για να υπάρξει ενημέρωση για τα ιατρικά τεχνολογικά προϊόντα. Ευχαριστώ. Και πάλι, ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο τριμερής διάλογος για τα medical devices, για τα τις ιατροπαραγωγικές ε, ε, συσκευές για τα ιατροπαραγωγικά προϊόντα και για τι διαδικασίε in vitro. το οποίο έλαβα από την ε, κυρία Μπέρα από την προηγούμενη θετία. Ξεκίνησε και αυτό δυναμικά με τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία και η Γκλένις Βέλμουτ από την Επιτροπή περιβάλλοντο, που είναι η καθήλυνα αρμόδια το κοιτάμε το θέμα αυτό και συμβάλαμε ως Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς σε μεγάλο βαθμό και προσπαθώ να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι που το εκτιμούν. Προχωρήσαμε ως τώρα σε κάποια μικρά θέματα. Καταφέραμε να περάσουμε και να προσπίσουμε την τοποθέτηση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ σε πολλά θέματα, αλλά η Λουξεμβουργιανή Προεδρία αποφάσισε στην παρούσα φάση μιας και τα πράγματα πηγαίνουν ε, πολύ αργά, να συμφωνήσουμε για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα υπό την Ολλανδική Προεδρία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να προσέξουν το θέμα αυτό, όσοι ενδιαφέρονται για τους τριμερούς διαλόγους, να το συζητήσουν μαζί μου και με τη Γραμματεία για να μπορέσουμε να λάβουμε τι ε, σημαντικέ και απαραίτητε πολιτικέ αποφάσει. Ε, Ω τώρα θα πρέπει να ομολογήσω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος με μεγάλη με ανοιχτό πνεύμα και επικοδομητική διάθεση αντιμετωπίζει τις απόψεις μας και στην προηγούμενη θητεία ε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος, άρα στην παρούσα φάση δεν έχω παρά στοιχεία να αναφέρω, αλλά για την ε, συμφωνία με το Συμβούλιο, ας είμαστε ρεαλιστές, δεν θα την πετύχουμε και τόσο γρήγορα. Είναι δύσκολο να συνοψίσουμε, γιατί αφενός ε, τα ιοτροφαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα in vitro, μέσω των δύο ε, οδηγιών, μετά το σκάνδαλο και μετά εμφυτεύματα στήθους, θα πρέπει να φροντίσουμε να τοποθετηθούμε καλύτερα στην αγορά. Από την άλλη, και οι υπουργοί το δήλωσαν αυτό, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε για το πώς θα, το πώς θα εξαιρέσουμε τα νοσοκομεία από το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας και σε τελική ανάλυση ε, κατέληξαν όλες οι ομάδες ότι αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον του ασθενούς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μια καλή λύση στο θέμα αυτό, αλλά ενδεχομένω, όπως σας είπα, αυτή η λύση να καθυστερήσει και λίγο. Ελπίζω με τον τρόπο λοιπόν αυτό, κυρία Πρόεδρε, να σας ε, παρουσίασα τα πιο σημαντικά στοιχεία του τριμερούς διαλόγου. Η πρόεδρο, θα ήθελε κανείς να θέσει και κάποιο θέμα, κάποια παρατήρηση, κάποια ερώτηση για το θέμα αυτό. Κάτι που αφορά ε, εμπορικά, μάλλον ζητήματα καταναλωτών και που εκφράστηκε προ εμένα ω ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία ότι όταν θα περάσει αυτό το νέο καθεστώ, τα υφιστάμενα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια, ενδεχομένω να καταστούν ε, παράνομα ή να χρειαστεί να περάσουν από μια νέα διαδικασία πιστοποίηση. και το ξέρουμε ότι οι καταναλωτέ πάντα θορυβούνται όταν ε, τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν ε, πλέον δεν είναι πιστοποιημένα και αναρωτιούνται γιατί Ιδιαίτερω αν κάποια από αυτά είναι βηματοδότες, ε, πρόσθετα κτλ. που τα χρησιμοποιούν επί σειρά ετών. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι θα γίνει με τις μεταβατικές αυτές φάσεις και πώς θα περάσουμε από το νέο, από το παλιό καθεστώς στο καινούριο. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό σήμερα, να έχετε υπόψη το πώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την μετάβαση των ασθενών, των καταναλωτών, γιατί ξέρω ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε σχέση με την αρχική πρόταση. Και αυτά συζητιούνται στους σήμερους διαλόγους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να σας δώσω οριστικές απαντήσεις σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια κάποια διάθεση και δημιουργείται η εντύπωση ότι με τα νέα πιστοποιητικά θα υπάρξει περισσότερη ασφάλεια. Νομίζω ότι δυστυχώς ε, δεν θα ισχύσει αυτό. Δεν ισχύει μάλλον αυτό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το εξή. Τα πιστοποιητικά που υπάρχουν να μπορούν να ελέγχονται ακριβώς κατά πόσον ισχύουν και κατά πόσον στέκουν. Να υπάρχει 100% εφαρμογή και υλοποίηση του ήδη φυστάμενου δικαίου και της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας. Το κατά πόσον τώρα χρειάζεται μια διαδικασία πιστοποίησης για περισσότερη ασφάλεια είναι αμφιλεγόμενο αλλά μέχρι εκεί υπάρχει μεγάλη συμφωνία και σύγκληση απόψεων μεταξύ των εισηγητών. Το Συμβούλιο, ωστόσο, ε, ακολουθεί μια πιο δύσκολη θέση. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε για να βρούμε μια λύση προκειμένου προ όφελο και προ το συμφέρον των ασθενών να μην επιβαρύνουμε με επιπλέον κόστο και διαδικασία πιστοποίηση προϊόντα τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν πρέπει να βελτιωθούν και σε τίποτα, μόνο θα κρυβίνουμε την όλη διαδικασία. Σίγουρα μου έχει μεταφερθεί αυτό το ζήτημα για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών και μετά υπάρχουν ζητήματα με την πιστοποίησή τους. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ. Σημείο για την διακυβέρνηση της αγορά αγοράς και ευρωπαϊκό εξάμεινο, η Κάθριν Στάλλον είναι συγγήτρια και εξέταση του σχεδίου έκθεση. Είναι μια έκθεση που εκπονούμε κάθε χρόνο. Γιατί σε έκθεση προόδου ανακοινώθηκε, δημοσιεύθηκε μάλλον στι 26 Νοεμβρίου. Όλοι λοιπόν είχατε δυνατότητα να τη δείτε. ιδίω σε ό,τι αφορά τι συστάσει για την Ευρωζώνη. που είχαν δημοσιευθεί μεταγενέστερα, τουλάχιστον αυτό λένε οι παρατηρήσει μου. Θα έχουμε μία σύντομη παρουσίαση τη ετήσια έκθεση προόδου με έμφαση, ιδιαίτερη έμφαση στην ενιαία αγορά. Πρώτα η συγγήτρια, και μετά Σαμπίν Βέιαντ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κάθριν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρίσταται σήμερα εδώ για να μας παρουσιάσει τις προτάσεις της για την ετήσια έκθεση προόδου. Εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω τη δική μου έκθεση για την διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του εξαμήνου του 2016. Όπως ξέρουμε, η ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά οικονομική ευημερία και για το παρόν και για το μέλλον. Και το, η δυναμική και η δυνατότητα που μα δίνει και θα μπορούσε να μα δώσει αυτή η ιστορική αγορά είναι ένα 3 ευρώ. Επομένω, λειτουργεί προ όφελο όλων μα. Αυτή τη στιγμή όμω υπάρχουν πολλά φράγματα και προσκόμματα, εμπόδια για την εσωτερική αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά κράτη-μέλη δεν υλοποιούν τι ε, αποφάσει τι οποίε έχουν προσυπογράψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω χρειάζεται και τα 28 κράτη-μέλη ε, και τη συνεργασία μεταξύ του. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η έκθεση για την ενιαία ε, διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς ε, στο πλαίσιο του εξαμήνου 2016. Αποτελεί τμήμα του, ενός πακέτου για τρεις κοινοβουλευτικές εκθέσεις που ε, αφορούν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2016. Οι άλλες δύο θα εξεταστούν από τις Επιτροπές Econ και EMPL. Έχουμε σπάσει την έκθεση σε τέσσερα σημεία ε, για κάθε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τρικής αγοράς ως ένα σημαντικό μέσο για την ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση ε, ε, η δυναμική και δυνατότητα δυνατότητα τη εσωτερικής που δεν έχουμε ακόμα εφαρμόσει, τα εφαρμοστικά μέσα, που αφορά τη συμμόρφωση και άλλα ζητήματα, αλλά είναι απαραίτητα για την ε, χρηστή διακυβέρνηση τη εσωτερική αγορά. Θεωρώ ότι απαιτείται ε, συντονισμό μάκρο- και μικροοικονομικών πολιτικών μαζί με το συντονισμό δημοσιονομικών πολιτικών ε, για να διαρθώσουμε καλύτερα την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Οι δυνατότητε που μα δίνει η εσωτερική αγορά έχει αναγνωριστεί πολλέ φορέ. Όμω, παρότι υπάρχουν συνεχώ εκκλήσει για, στην ετήσια έκθεση προόδου και στι ειδικέ αναχώρα συστάσει δεν έχει υπάρξει ουσιαστικά πρόοδο. Μεταξύ του 12 και του 2013 περίπου 10% μόνο των ειδικών αναχώρα συστάσεων έχουν υλοποιηθεί πλήρω ή σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη. Για να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα, η πρόοδο σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά στα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία το να συμπεριλάβουμε τον πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, Παρακολουθώντα δηλαδή και την ευημερία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, ιεραρχώντα προτεραιότητε, κυρίω ό,τι αφορά την απασχόληση, αυτό θα ήταν μια καλή πρόοδο. Πρέπει να έχουμε μια εύρωστη βάση δεδομένων με ποσοτικού και ποιοτικού δείκτε, σημεία αναφορά, αναθεώρηση ομοτήμων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ε, ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά. Θα αυξάνεται η ψηφιοποίηση και η διαλειτουργικότητα. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικέ μα να είναι στραμμένε προ το μέλλον και να έχουν ένα μεταμορφωτική συνέπεια και αντίκτυπο στι ζωέ των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί πλέον ε, γίνεται πιο δυσδιάκριτη η διαφορά μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε όλους ε, τους πελάτες να κάνουν συναλλαγές ε, στο διαδίκτυο και τα άλλα υλικά και προϊόντα και αγαθά μάλλον ε, αναλαμβάνουν μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τα υλικά. Αυτή είναι λοιπόν μια κατάλληλη προσέγγιση για το μέλλον. Η εμβάθυνση τη τουρκική αγορά σε όλου του τομεί πολιτική δεν πρόκειται να επιτευχθεί εάν ε, η στρατηγική αυτή ε, την εξετάσουμε από μόνη τη. Πρέπει να συνοδεύεται και να υπάρχει δανεισμό και με άλλες πολιτικές για την Ενεργειακή Ένωση, την Ένωση Κεφαλαγορών ε, και το πακέτο της κυκλικής οικονομίας. Βεβαίω πρέπει να υπάρχουν μικρο- και μακροοικονομικές πολιτικές, ε, έγκαιρη και κατάλληλη εφαρμογή όλων αυτών των πολιτικών από όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι απαραίτητη προπόθεση για την ε, ευημερία και την κατάλληλη λειτουργία τη εσωτερική αγοράς. Δεν ήταν εύκολη δουλειά αυτή η έκθεση. Το ξέρετε και πολλοί από εσά που ήσασταν εισηγητέ ότι είναι δύσκολο κάποιο ε, να ε, αντιμετωπίσει επαρκώ ε, όλου αυτού του τομεί πολιτική και τα επιμέρου κομμάτια τη ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, την οδηγία περιπηρεσιών και άλλα τέτοια παραδείγματα. Κάτι άλλο το οποίο είναι δύσκολο. Ναι, με ενθουσιάζει ιδιαίτερα η ενιαία αγορά. Όμω, με λυπεί το γεγονό ότι η έκθεση έπρεπε να οριστικοποιηθεί και να σταλεί για μετάφραση πριν από την δημοσίευση τη αιτήσια έκθεση πρόοδου. Γι' αυτό είναι σημαντικό που είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω προσπάθησα να δυσφαλίσω ότι τα προηγούμενα στοιχεία θα ενσωματώνονται καλύτερα στην τελική εκδοχή ε, τη έκθεσή μου πριν περάσει στην ε, Επιτροπή στι 25 Ιανουαρίου. Περιμένω λοιπόν να ακούσουμε ενδιαφέρον ε, την παρουσίαση της Κομισιόν. Ξέρω ότι έχουμε μία ε, συνεδρίαση των σκιωδών αύριο και μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλονται τροπολογίες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και προσβλέπω και σε περαιτέρω συζητήσεις και με τους σκιώδεις στο εγγυσμένο. Ευχαριστώ. Do we want to take a round from... Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις πρώτα. Or, Mr. Zulik, as Dan, are you... Or can we listen to the Commission first? Ίσως η Επιτροπή πρώτα, περιμένοντας τον Άνταμ. He's here. Welcome. Um, so we started already and the rapporteur has... Καλώς ήρθατε, η συγγήτρια παρουσίασε την έκθεσή της. Okay, Dan. Thank you, Chair. I'll take advantage of this elevation. Λοιπόν, θα εκμεταλλευτώ την τιμητική για την ομάδα μου. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Στάιλα για την ε, πρότασή της είναι μια θετική πρόταση στις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της ε, ενιαίας αγοράς. Ο κύριος Σούλικ μένει στους δίκτες της ενιαίας αγοράς και στην ένταξη των δικτών αυτών στις διαδικασίες η κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πραγματικό κίνητρο για την ανάπτυξη, δεν προϋποθέτει δημόσιες επενδύσεις και είναι μία μέθοδος βελτίωσης άνευ κόστους. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν με τις προτάσεις αυτές και εγώ προσωπικά. Ο κύριος Σούλικ ταυτόχρονα και το σύνολο της ομάδας νομίζω θεωρεί ότι η βασική δραστηριότητα της Ένωσης είναι ακριβώς η ενιαία αγορά. Υπάρχουν δύο τομείς τους οποίους πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, ο κ. Σούλεκ. Καταρχάς, σε σχέση με τον τρόπο λήψης ε, αποφάσεων είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να, ε, να αποδυναμώσει ε, τον δυναμισμό των περιφερειών της Ευρώπης και δεν θα πρέπει εμείς να συγχαίουμε τη μακροοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τα επιμέρους μέτρα τα τομεακά βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Θα έχουμε κάποια προβλήματα και με την έκκληση για αύξηση δημοσίων δαπανών στον τομέα της ICT και θα θέλαμε η συγγήτρια να είναι πιο ξεκάθαρη ακριβώς με την πρότασή της. Κατά τα άλλα δεν έχω κάτι να προσθέσω εκ μέρους του κυρίου Σούλεκ. Ευχαριστώ Σάντφιλντ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Τα αεροπλάνα δυστυχώς καθυστερούν. Χαίρομαι λοιπόν που προχωράμε με την υπόθεση αυτή. Διάβασα την πρόταση ε, με μεγάλη ικανοποίηση θα έλεγα και θα πω ειλικρινώς ότι υπάρχουν πολλά σημεία στην γνωμοδότηση με τα οποία θα συμφωνήσω πλήρως. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά να προσθέσω. Λίγα ε, παρατηρήσεις όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω. Επαναλαμβάνω όμως ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι κεφαλαιόδου σημασίας δεν αντιμετωπίζεται πάντα σαν τέτοιο στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι στην επόμενη φάση η θέση μας ε, δεν είναι πάρα πολύ ε, ευτυχής. Ένας από τους λόγους είναι η ατελής λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η αποτυχία μας να κατανοήσουμε την σημασία της ενιαίας αγοράς. Και εάν δεν σεβαστούμε τις αρχές που θα επιτρέψουν το streamlining της αγοράς, τότε η ανταγωνιστικότητά μας θα υπονομευθεί ακόμα περισσότερο. αν θέλουμε να παραμείνουμε μια οικονομική υπερδύναμη και αν συγκρίνουμε το τι κάνουν άλλες οικονομικές ε, ε, υπερδυνάμεις θα δούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία έχουν αγορές οι οποίες σε εσωτερικό επίπεδο είναι ιδιαίτερο συνεκτικές και η ζήτηση στις αγορές αυτές δεν περιορίζεται σε καμία περίπτωση από εσωτερικά εμπόδια. Θα πρέπει λοιπόν καλούμεθα να ανταγωνιστούμε με τις αγορές αυτές, αλλά δυστυχώς έχουμε προβλήματα ακόμα στην δική μας εσωτερική αγορά. χάνουμε εκατομμύρια καταναλωτές και έτσι ε, μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και μειώνονται και οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο επιθυμητό που είναι η ευμάρεια των πολιτών. Απαιτείται λοιπόν μια σωστά λειτουργούσα εσωτερική αγορά και μια αγορά με τέτοιου είδους εμπόδια δεν μπορεί να προοδεύσει δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα σωστό κλίμα για τη δημιουργία και τη λειτουργία των μικρομεσαίων. Οι μικρομεσαίες θα πρέπει να δαπανούν τεράστια ποσά ε, ενέργειας αντιμετωπίζοντας γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία λειτουργούν αντί αναπτυξιακά. Κάποιες από τις ε, μικρομεσαίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κινητικές, αναζητούν ευκαιρίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό λοιπόν θα συμφωνήσω με τον εισηγητή, ότι πρέπει να στην εισηγήτρια μάλλον, ότι βασικός μας στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Πέραν τούτου, ciągle Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποσύρουμε από τη μέση τα εμπόδια αυτά. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Σαν παράδειγμα υπάρχουν ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες ε, για τις ε, ελεγχόμενες ε, ειδικότητες και με ακριβώς αυτές τις διαφορετικές αναχώρα ρυθμίσεις η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάποιος ο οποίος ασκεί το επάγγελμά του σε μία χώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι έστω και προσωρινά σε μία άλλη. Μιλάμε για το λεγόμενο διαβατήριο των υπηρεσιών. Μα γιατί αναζητούμε μια τέτοια λύση. Γιατί να μην αναγνωρίσουμε ότι τα επαγγέλματα, εν πάση περιπτώσει, που αναγνωρίζονται σε μία χώρα, θα πρέπει η αναγνώριση αυτή να ισχύει και στην άλλη. Λοιπόν, αυτά χοντρικά. Powodować, by także e, komisje Parlamentu Europejskiego Σημασία λοιπόν περισσότερη στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει και οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές να αντιμετωπίσουν το θέμα με την ίδια προτεραιότητα. Thank you. Um, I'm speaking on behalf of Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ ονόματο του συναδέλφου είμαι Σκιώδη. Ο κύριο Γκόμπα, λοιπόν, ευχαριστεί ε, την εισηγήτρια για το σχέδιο νομοδότηση. Είναι εξαιρετική δουλειά τη κυρία εισηγήτρια, θεωρεί ο κ. Κόγκα, και συμφωνεί με τι προτάσει τη. Για την ομάδα Alde, είναι προφανές ότι η εσωτερική αγορά είναι εξαιρετικά πολύτιμη για την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, ιδίω τώρα που η εσωτερική αγορά έχει να αντιμετωπίσει και την ψηφιοποίηση. Ο κ. Γκόκα συμφωνεί πλήρως με την εισηγήτρια για την ανάγκη να επικεντρωθούμε περισσότερο στην εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την αναγκαιότητα ανάπτυξη αναλυτικών ε, μέσων για την ε, μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων Υπάρχει έλλειψη τη υλοποίηση, ανεπαρκή υλοποίηση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε σε διαδικασίε παραβάσει. Ο κ. Βόγκα θεωρεί ότι είναι κρίμα που τα σημεία επαφή προϊόντων δεν λειτουργούν ω ενιαία θηρίδα για σημαντικά ζητήματα τη ενέργεια αγορά και θα πρέπει να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ενεργήσει περισσότερο σε ό,τι αφορά την αρχή τη αμοιβή αναγνώριση, που είναι κρίσιμη σημασία στοιχείο η λήψη εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο κ. Γκόγκα θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει την ε, δυναμική τη ε, οικονομία με βάση τη συνεργασία και για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων για να διαμορφωθούν οι κατάλληλε συνθήκε να αναπτυχθεί η αγορά πρέπει να έχουμε νέα νομοθεσία για την εποπτεία της αγοράς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν έχει κάνει αρκετά σε αυτό το τομέα μέχρι τώρα. Θεωρεί ότι η ανταγωνιστική ενιαία αγορά στην Ευρώπη για τον 21ο αιώνα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μεταρρυθμίσεις ό,τι αφορά ε, τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σε πολλά κράτη-μέλη ε, καταδεικνύει ακριβώς την αναγκαιότητα φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων. Συμφωνεί με τις δυνατότητες ε, των ηλεκτρονικών προμηθειών, όμως ε, επισημαίνει και την ανάγκη άμεσης ε, και πλήρους εφαρμογής της, οδηγίας, της σχετικής οδηγίας σε όλα τα κρατημέλη. Και τέλος θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ε, έναν δημόσιο τομέα με λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερε επιδόσει. Βάσει και τη νομοθεσία ISA 2, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο δημόσιο τομέα είναι σε θέση ε, να συνεργάζεται με άλλου δημόσιου τομεί σε διασυνορικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Εντάξει, από πλευρά ΓΟΕ, κύριο Ζούμπα. Δεν είναι εδώ. Και για τους πράσινους, Πασκάλ Ντογάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω αφενός να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και εγώ θεωρώ ότι συμμεριζόμαστε πολλές από τις απόψεις της. Επομένω, ε, πρόκειται για σημαντική πρόοδο από αυτή τη σκοπιά. Τώρα, μερικές παρατηρήσεις μόνο επί της ουσίας. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν πρέπει να αποτελεί μόνο δημοσιονομικό εγχείρημα. Πρέπει να καταφέρουμε να υπάρξει αυτή η ολοκλήρωση και να υπάρχει ένα ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος ε, συμφερόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευρωπαϊκός χώρος δημόσιου συμφέροντος παρόλε τι διαδικασίε που έχουμε στο Κοινοβούλιο και τα καθεξή, νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζουμε όλα τα σημεία προβληματική που τίθενται. Για παράδειγμα, το ζήτημα τη κυκλική οικονομία είναι σημαντικό θέμα, γιατί μπορεί να αποτελεί και μία από τι δυνατότητε ε, που έχει η Ευρώπη ε, για να εισέλθει στον 21ο αιώνα ε, ανακυκλώνοντας και τους πόρους της και επανατοποθετώντας και τις δυνατότητες που έχει είναι λοιπόν ε, αυτή η δυνατότητα που έχουμε για την ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τις δημοσιοπρομήθειες κατανοώ ότι πρέπει να το εξετάσουμε και από τη σκοπιά. Πράγματι, ε, οι δημόσιε δαπάνε αποτελούν περίπου 20% των επενδύσεων στην Ευρώπη. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντική διάσταση και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε την ψηφιακή οικονομία χωρίς ε, να λάβουμε υπόψη και τις επενδύσεις στην έρευνα ή και αλλού που ε, κατά κύριο λόγο είναι δημόσιες επενδύσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν που το αναφέρουμε και που το αναφέρετε κι εσείς και συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Τώρα για να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία στην έκθεση βλέπουμε, για παράδειγμα, την ε, άρση των εμποδίων που και εμείς επιθυμούμε βεβαίως. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα ζητήματα ε, του ανταγωνισμού και μεταξύ κρατών. Σε ό,τι αφορά ας πούμε, τις αρχές εποπτείας της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι υπάρχει μια, ένας αναπαρκής έλεγχος ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. δεν θέλω να μπούμε σε αντιπαράθεση, αλλά ε, ε, ας πούμε η υπόθεση Volkswagen, αλλά και για άλλες εταιρείες ισχύει αυτό, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ των αρχών εποπτείας, των κρατών μελών και των επιχειρήσεων αυτών. Επομένως υπάρχει σημαντική ανεπάρκεια έλλειψη ε, υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος στην Ευρώπη. Θα ήθελα να επιμείνετε εδώ για να υπάρχουν πραγματικά ε, Ευρωπαϊκέ αρχέ εποπτεία που θα υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Σβάπ. και δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι σκιώδη συζητητή. Ε, παρ' όλα αυτά χαίρομαι που ε, διάβασα την έκθεση της συναδέλφου και όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι συμφωνώ με πάρα πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται αλλά ακριβώς επειδή έχουμε μαζί μας σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο Καταρχάς, να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος Σάινφελτ ως προς το περιεχόμενο. Σε βάθος χρόνου θα διατηρήσουμε την ευημερία στην Ευρώπη μόνο αν έχουμε ανταγωνιστικότητα και μάλιστα σε διεθνέ προσκήνιο. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας. Η ερώτηση που έχω να κάνω, κυρία Στάιλερ, είναι το εξή. Από πού, σε τι είναι διαφορετική η έκθεση για την ε, διακυβέρνηση της ενίας ε, αγορά σε σχέση με τις υπόλοιπες σχετικές ε, εκθέσεις. Μιλάτε για τη στρατηγική, Στην συνάδελφος μιλά για τη στρατηγική, για την ενιαία αγορά. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν ε, διαφορετικά σημεία εστίασης, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ε, σε τι έγκυται αυτή η διαφορά. Υπάρχει και το ευρωπαϊκό εξάμεινο και πάντα σε τέτοια ζητήματα Επικεντρωνόμαστε στα ζητήματα που εμποτίζουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και στις συστάσεις αναχώρα. Και οι σοσιαλδημοκράτες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση των ζητημάτων αυτών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και πράσινη πράσινοι επίσης και στο θέμα της ε, εσωτερικής αγοράς θεωρώ ότι το, οι σαν χώρα αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα, αλλά αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και επειδή έχουμε εδώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω ότι θα πρέπει από κοινού να θέσουμε το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο ρόλος ε, της ενιαίας αγοράς, τι αποτέλεσμα θα πρέπει να έχουν αν συζητάμε μία φορά το χρόνο για την ενιαία αγορά και η γνωμοδότηση αποστέλλεται απλά προς την αρμόδια επιτροπή. Ε, ας μην το κάνουμε καθόλου. Να ξέρουμε όμως ποιο σκοπό επιδιώκουμε με την έκθεση αυτή. Γιατί τα στα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και περίπλοκα. Και γι' αυτό πιστεύω αυτό δεν θα είναι δίκαιο καν για τη συνάδελφο. Και αν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα κάποιος άλλος ε, να πάρει το λόγο πριν την Επιτροπή. Η κυρία Βέντ, συντονίστρια πολιτικής, θα κάνει μία σύντομη παρουσίαση για την έρευνα για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Στάιλερ, αγαπητά μέλη. Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη και θα συγκεντρώσω την προσοχή μου στους τομείς ε, που ενδιαφέρουν και την Επιτροπή σας, που είναι αρμοδιότητά σας και ταυτόχρονα θα δώσω κάποιες πρώτες απαντήσεις στις ερωτήσεις του κ. Σφάρτς. Δημοσιεύσαμε το πακέτο μας στο τέλος Νοεμβρίου, είναι η αρχή του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το πακέτο αυτό συνίσταται από την έκθεση για το 2016, έκθεση ανάπτυξης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο ε, μεμονωμένων κρατών μελών στον οικονομικό και νομισματικό τομέα. Είναι το πρώτο βήμα το οποίο γίνεται επίσης στην ε, ανείχνευση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη στο εσωτερικό των κρατών μελών. Αναλύουμε επίσης και την κατάσταση της απασχόλησης στα διάφορα κράτη-μέλη και όπως είπε η Πρόεδρος στην αρχή έχουμε επίσης προχωρήσει και στις συστάσεις για την Ευρωζώνη τονίζοντας την αλληλοεξάρτηση και την υποχρεωτική σύγκληση των χωρών που συμμερίζονται, που μοιράζονται μάλλον το ευρώ. Στα πλαίσια λοιπόν της έκθεσης για την ανάπτυξη το 16 προσπαθούμε να φτιάξουμε την ιεραρχία των πολιτικών σύγκλησης. Και φυσικά εδώ τίθενται και τα θέματα της ενιαίας αγοράς και της στρατηγικής για τη βελτίωσή της. Η ετήσια έκθεση λέγει ότι θα πρέπει εμείς να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα όθηση των χαμηλών τιμών των πρώτων υλών και της χαμηλής ισοτιμίας του ευρώ συν της ε, ε, διευκολυντικές νομισματικές πολιτικές έτσι ώστε να προωθήσουμε την οικονομία. Δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε μιας και δεν έχουμε στην παρούσα φάση άμεση πίεση αλλά να δημιουργήσουμε πόρους για το μέλλον. Αν εξετάσει κανείς την έρευνα για το 16 θα δει ότι υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός συνέχεια σε σχέση με το 2015 στον τομέα της ε, της τρίγωνης πολιτικής, δηλαδή επενδύσεις, διαφθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές. Υποστηρίζω ότι οι δύο από τις τρεις καλύπτουν τις δικές σας αρμοδιότητες. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η έκθεση για το 16 υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο τη σημασία του τομέα των επενδύσεων. Τον τομέα των επενδύσεων και χάρη ακριβώς στην γρήγορη αντιμετώπιση του θέματος στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Έχουμε προχωρήσει με το πλάνο για τις στρατηγικές επενδύσεις του Προέδρου. Έχουμε μπει στις διαδικασίες χρηματοδότησης. Ο δεύτερο πυλώνα που είναι ο εντοπισμός των προσχρηματοδότηση προγραμμάτων και τρίτον να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε τα διακανονιστικά θεσμικά εμπόδια. Αυτά τα εξετάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενιαία αγορά, εφαρμογή κανόνων, συμπεριφορές, αποδοχή, αλλά και προσπαθούμε να δούμε επίσης και σε εθνικό επίπεδο τι γίνεται και όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν μέσω και της εναρμόνισης. Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε με διαφορετικό τρόπο την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν όμως θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ως εκ τούτου θέλουμε να είμαστε σε συζήτηση μαζί τους για τα θέματα αυτά. Ένα παράδειγμα είναι οι δημόσιες προμήθειες. Η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά ανεπαρκής αφέ αυτής, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να ωφεληθούν πλήρως από τις ανταγωνιστικές ελεύθερες αγορές. Θα πρέπει λοιπόν και σε σχέση με την ενιαία αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και το εξάμεινο για να προχωρήσουμε σε μία μορφή διαλόγου με τα κράτη-μέλη. Παράδειγμα ήταν οι δημόσιες προμήθειες. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους υπάρχουν εθνικές ρυθμίσεις για θεμητούς πολιτικούς λόγους. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς στους οποίους τίθεται το ερώτημα εάν οι ρυθμίσεις οι εθνικές είναι οι λιγότερο στρεβλωτικές. Εδώ τίθεται λοιπόν το θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς και ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε πει πέρυσι, τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Εδώ πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με τα κράτη-μέλη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το 2016. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να εντάξουμε τα προϊόντα μας καλύτερα στις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγορών και στις παγκόσμιες αλυσίδες συναλλαγών η πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρούσα φάση διευκρινίζει ότι ε, πρέπει να ενισχυθεί ο μικροοικονομικός πυλώνας. Μιλήσαμε για τη μακροοικονομία, για τα δημοσιονομικά, αλλά και το μικροοικονομικό είναι ένα τομέας στον οποίο ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Αυτό θα μας απασχολήσει για το 16. Τι εννοούμε με αυτό. Όπως φαίνεται και στα πλαίσια της έκθεσης για την ανάπτυξη, έχουμε κυκλοφορήσει μια, ένα εσωτερικό έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στοιχεία ανακράτος μέλος για τα βασικά εμπόδια στις επενδύσεις όπως βγήκαν από τις επαφές που είχαμε με τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα. Υπάρχουν χώρες λοιπόν οι οποίες θέλουν να εμβαθύνουν το διάλογο μαζί μας και την ανάλυση μας έτσι ώστε να υπάρξουν καλύτερες προτάσεις τον μήνα Φεβρουάριο όταν δημοσιεύσουμε τις country reports, τις εκθέσεις αναχώρα. Αυτή είναι η βάση για το επόμενο βήμα στα πλαίσια του εξαμήνου που είναι οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Φυσικά και στην παρούσα φάση δεν είμαι σε θέση να σας πω εγώ ποιες θα είναι και σε ποια σημεία θα επιμείνουν οι συστάσεις αναχώρα. Γνωρίζετε ότι οι κύριοι κύριοι Γιούνκερ Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι επίτροποι αποφάσισαν πέρυσι οι συστάσεις αυτές να γίνουν πλέον με τρόπο πολύ πιο ευθυγραμμισμένο από ό,τι στο παρελθόν και πολύ πιο συγκεκριμένο. Αυτό όμως δεν ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι πολύ ευρύτερο, έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια έχει ένα ολόκληρο πλάτος δυνατότητας ανάλυσης και πρέπει να το διασώσουμε και τα προβλήματα της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνονται σε αυτό. Και τα βλέπω αυτά και στην έκθεση της κυρίας Στάιλα. Ως εκ τούτου λοιπόν και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει σύνδεσμος ισχυρός ανάμεσα στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επί τη βάση αυτής της ανάλυσης θα δημοσιεύσουμε τις αναλυτικές παρατηρήσεις μας αναχώρα τον μήνα Φεβρουάριο και θα κάνουμε τις απαιτούμενες προτάσεις. Ελπίζουμε ότι και επί τη βάση της θεματολογικής ανάλυσης την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η Επιτροπή σας θα εξετάσει θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη γκάμα υλικών και αναλύσεων οι οποίες μπορεί να προωθηθούν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αντικείμενο πλήρους εκμετάλλευσης. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ιδέες στην πρόταση εκθέσεως ε, για να ενισχυθεί ακριβώς ε, ο μικροοικονομικός, ε, η μικροοικονομική κλίμακα αν θέλετε και να αυξηθεί και να εμβαθυνθεί ο διάλογος με τα κράτη-μέλη και εμείς είμεθα ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για την συνεχιζόμενη εμπλοκή της δικής σας Επιτροπής. Δεν έχω κάτι άλλο να πω στην παρούσα φάση, περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση. Και πρωτού επαναληφθούμε στο, στη συγκεκριά, θέλει κανείς το λόγο από τα μέλη που μόλις κατέφτασαν, η κυρία Γκέπαρτ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησε η πτήση μου και γι' αυτό δεν μπόρεσα να έρθω στην ώρα μου αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το έργο για τα εξάμεινα που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα ομολογήσω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές συστάσεις, αλλά ρωτιέμαι σε τελική ανάλυση τι αποτέλεσμα βγαίνει από όλο αυτό το έργο, γιατί από ένα σημείο και πέρα ειλικρινά δεν έχω όρεξη να δουλέψω, αν δεν υπάρχει και κάποια α, συγκεκριμένη κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πολλά ακούμε, πολλά λέμε, και από τα κράτη-μέλη, αλλά λίγα γίνονται. Και ως εκ τούτου κατανοώ, κατανοώ το γεγονός ότι πολλοί πολίτες αναρωτιούνται πλέον για το όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Και νομίζω ότι προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται η κυρία Στάιλερ και ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ ε, συγκεκριμένες συστάσεις, όχι μόνο αναλύσεις, αλλά το τι θα πρέπει να κάνουμε για να υπάρχει πραγματικά επιτυχία και ανάπτυξη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θέσεις ε, εργασίας ε, και να ανοίξουν και συγκεκριμένες προοπτικές για τον κόσμο που κατά τα άλλα ενδεχομένω να μην έχει κάποια ευκαιρία. Και νομίζω ότι η δική μας η Επιτροπή στο συγκεκριμένο σημείο έχει πολλά να προσφέρει. Και αυτή είναι η δεύτερη διάσταση η οποία με ενοχλεί και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι προφανώς και δεν θέλω να εξαιρέσω οποιαδήποτε ομάδα ότι δεν αναγνωρίζεται όπως θα έπρεπε και η σημασία της ε, Επιτροπής ε, ε, προστασία του καταναλωτή και τη εσωτερική αγορά. Δεν είναι μόνο το θέμα τα χρήματα. Το θέμα είναι ποια είναι η βάση. Υπάρχει κάποια κοινή βάση. Ή ο καθένα κάνει ό,τι νομίζει και στη τελική ανάλυση πάλι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στα κατεπήγοντα ευρωπαϊκά ζητήματα τη ανεργία, τη γενικότερη κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του τι θέλουμε στο μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεξή. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ και για τη δική μας επιτροπή, αλλά νομίζω ότι θα το πετύχουμε σε κάθε περίπτωση με την κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πολύ. Αναπτύσσουμε σίγουρα ε, ένα πολύ ισχυρό προφίλ για την Επιτροπή μας. Είμαστε πιο μικρές επιτροπές, αλλά φωνάζουμε πιο δυνατά από όλους. Η Κάτριν να πάρει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, μπορεί να είμαστε μικρή επιτροπή, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχολούμαστε με την ενιαία αγορά, με τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολλές απόψεις. Ε, μίλησε ο Ντάνιελ για θέματα που έχουν να κάνουν με το ΕΣΤΗ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τα της στρατηγικής για την ενιαία αγορά. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα μπει στην ε, ενιαία αγορά. Το 17% ε, του ICT ε, δαπανάται στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Αυτό για να τονίσουμε τη σημασία του ICT. Για αυτό που αναφέρθηκε για την ε, κατάργηση των φραγμάων Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Πώς ε, τα άτομα που έχουν ε, διπλή διπλές ικανότητες που θα μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν Ξέρω ότι εκπροσωπείται επίση συνάδελφο τον κ. Κόγκαρα το θέμα για την ψηφιοποίηση που αναφέρατε. Είναι πάρα πολύ ουσιώδες και είναι σημαντικό που το τονίσατε. Επίσης, αυτό που είπε ο κ. Ντοράν για την κυκλική οικονομία. Ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε από την άποψη αυτή έχει να κάνει με την ε, γενικότερη επισκόπηση του πώς λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Όλη αυτή η σύνδεσμοι είναι σημαντική. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τρία σημεία που ανέφερε, τα τρία σημεία του τριγώνου για τις επενδύσεις, τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις και το καθεξής. Και στο τέλος που είπε και η κυρία Γκέπχαρτ για τις προοπτικές του πώς θα λειτουργήσει η Ένωση. Όπως σας είπα στον πυρήνα μας, έχουμε την εύρυθμα λειτουργούσα αγορά. Θα πρέπει όλα αυτά να μπουν πιο πολύ στο εξάμεινο και νομίζω ότι όλα τα στοιχεία αυτά από κοινού τονίζουν τη σημασία της ενιαίας αγοράς και έτσι οδηγούμαστε και πάλι σε αυτά που είπε η κυρία Ιγκεπχάρτ, γιατί δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο, αλλά και να έχουμε συγκεκριμένες πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση των σκηνοδών. Προθεσμία για τι ε, τροπολογίε, είναι η 16η Δεκεμβρίου, 25 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε που είναι και η ημέρα ενός Φιλανδού ποιητή. And then you'll buy everyone. Και μετά θα μας κεράσετε όλους ένα whisky. Και χάγκης βεβαίως. Okay. Um, it sounds, sounds to me as if they're making some good progress. It's also sound... Εντάξει, μου φαίνεται ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος και από ό,τι είπατε και εσεί θέλετε και προτίθεστε να υποβάλλετε από μόνοι σα τροπολογίες το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ συχνά εξαιρετικά χρήσιμο όταν μπορεί ο εισηγητής εκ των προτέρων να αποστέλει τις τροπολογίες ε, και στους κοιόδης για να υπάρχει μια συνεργασία και εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα μερικά λεπτά περιθώριο και ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το επόμενο σημείο. Ας ε, περιμένουμε λοιπόν 10 λεπτά για να ξεκινήσουμε στις 4 ε, και 20. Διάλειμμα 13 λεπτών, λοιπόν. Εκτός και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Όχι. So the Commission um, is here, but the person who was going to be presenting is not yet here. Είναι εδώ λοιπόν ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι το άτομο που θα κάνει παρουσίαση. Και επειδή είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, θα περιμένουμε.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 Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άνω των 20 μελών από πάρα πολλές χώρες και από πολλές πολιτικές ομάδες. Ο βοηθός γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έπρεπε να είναι παρόν. Μου είπαν ότι έρχεται. Θα μπορούσαμε ίσως να ζητήσουμε από κάποιον άλλο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Λόγω της σοβαρότητας όμως ε, του θέματος και, της, ε, ε, του ενδιαφέροντος των μελών θα πρέπει να περιμένουμε τον βοηθό γενικό διευθυντή έτσι ώστε να ακούσουμε άμεσα τη γνώμη μου. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν είναι εδώ, είμαστε ίσως πέντε λεπτά πριν από το πρόγραμμα. we were πριν 10 λεπτά μου είπαν ότι θα ήταν εδώ σε 2 λεπτά. Έπαθε τίποτα. So, um, Κυρίες και κύριοι, μίλησα με τους δανειστές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέσας διάταξης, γιατί θα ήθελαν να ακούσουμε την παρουσίαση του αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλησαν λοιπόν να αλλάξουμε τη σειρά των θεμάτων της μέσας διάταξης. αλλά δεν είναι εδώ. So we will continue to wait. Θα περιμένουμε κι άλλο λοιπόν. Um, okay, so we're going to move on to an item. Λοιπόν, θα περάσουμε στο σημείο 7 της ημίσης διάταξης, παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια πρόταση οδηγίας για τον έλεγχο επί της απόκτησης και κατοχής ε, όπλων. Η λεγόμενη οδηγία προβολών όπλων ήρθε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής κ. Δελσάου. Πάντα σας ζητούμε να φτάνετε στην ώρα σας, γιατί ήταν πολλά και τα μέλη της Επιτροπής ε, παρόντα. Ε, από το 1991 υπάρχει ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία και το 2008 είχε αναθεωρηθεί από την Επιτροπή μας και ο προκάτοχος μου ήταν ένας από τους συγητές. Η αναθεώρηση περιλάμβανε και έναν εφαρμοστικό κανονισμό για να διασφαλίσουμε ε, την, ε, τον κατάλληλο παροπλισμό των ε, όπλων αυτών όταν ο παροπλισμός είναι απαραίτητος. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο που αυτός ο εφαρμοστικός κανονισμός μας έχει πάρει τόσο καιρό να τον συμφωνήσουμε, αλλά από ό,τι μαθαίνω εγκρίθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει και επέβαλε αυτή την πρόταση και μόλις το έμαθα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει στην Επιτροπή μας ε, και να την παρουσιάσει το στοματώρο δυνατόν. Ξέρουμε ότι η πρόταση περιλαμβάνει στοιχεία που θα βελτιώσουν ε, ε, την ανταλλαγή δεδομένων στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την καλύτερη ιχνηλάτηση αυτών των όπλων. Και ξέρω ότι υπάρχουν και σημεία προβληματισμού από το ευρύ κοινό για συγκεκριμένα τμήματα της διατύπωσης. Και γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Και ήθελα να επενθυμίσω και το ευρύτατο κοινό ότι είναι ο ρόλος της Επιτροπής αυτή, αλλά και γενικότερα των κοινοβουλευτικών επιτροπών, να υποβάλουν τροπολογίες ως προς τη διατύπωση. Αυτό συμβαίνει για κάθε νομοθετική πρόταση. Δεν είναι τελική δηλαδή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως ότου υποβληθούν και ψηφιστούν τροπολογίες από τις Επιτροπές. Και γι' αυτό είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχουν παραθυράκια, κενά, ελλείψεις. Παράλληλα, θα πρέπει μαζί με τη νέα νομοθετική πράξη να υπάρχει κατάλληλη αντιμετώπιση και των παράνομων πυροβολών όπλων. Και την περασμένη φορά που είχε υποβάλει η Κομισιόν πρόταση, εξέταζε ε, τα παράνομα όπλα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντελουσάου για να μας ε, παρουσιάσει την πρόταση. Και ξέρω ότι είναι αρκετοί οι συνάδελφοι, αρκετοί βουλευτέ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Του καλώ λοιπόν να ζητήσουν να μπουν στον κατάλογο μελετών. Κύριε Σάιντελ Σάου, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, λυπάμαι για την καθυστέρηση. Υπήρχε σοβαρό λόγο, σα διαβεβαιώ, αλλά και πάλι ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν, είναι, δεν μπορεί να γίνει δεκτή μια τέτοια στάση. Δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω το πλαίσιο και το υπόβαθρο, κατανοείτε την σοβαρότητα του ζητήματος και πόσο σύνθετο είναι αυτό το ζήτημα. Κατανοείτε λοιπόν το υπόβαθρο. Γιατί υποβάλλουμε αυτή την πρόταση. Θέλω να είμαι σαφής. Με την πρότασή μα δεν θέλουμε να λύσουμε όλα τα ζητήματα που συνδέονται με το θέμα των πυροβολών όπλων. Σε αυτό το κείμενο δεν επικεντρωνόμαστε στο παράνομο εμπόριο όπλων. Και όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Ασφαλείας που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου γίνεται προσπάθεια να αποτελέσει απάντηση στο μεγαλύτερο ζήτημα των παράνομων όπλων. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα που μας αφορά σήμερα, παρότι είναι εξαιρετικά σημαντικό βεβαίω. Τα μέτρα που προτείνουμε βασίζονται σε τρεις μελέτες που έχουν εκπονηθεί από συμβούλους και έχουμε εκπονήσει μια έκθεση της Επιτροπής που απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και η έκθεση αυτή αποτελεί αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας πυροβολών όπλων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Μόνιμη Διεθνή Επιτροπή για τα στοιχεία που μας έδωσαν και την εμπρογνωμοσύνη που μας έδωσαν για τα μικρά όπλα. Ποιες είναι οι πέντε βασικές αλλαγές που προτείνουμε να εισαγάγουμε στην οδηγία. Πρώτη σημαντική τροποποίηση αφορά τις κατηγορίες των πυροβολών όπλων. Θέλω να είμαι εξαιρετικά σαφής και σε αντίθεση με όσα έχω δει στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, ορισμένες αντιδράσεις. Εμείς δεν έχουμε ως στόχο να απαγορεύσουμε όλα τα ημιαυτόματα όπλα ε, και τη χρήση τους για τους ε, πολίτες. Σε ό,τι αφορά τα ημιαυτόματα όπλα. Θέλουμε να απαγορεύσουμε μόνο δύο κατηγορίες όπλων που έχουν ε, θεωρηθεί πιθανώς επικίνδυνα. Πρώτα τα αυτόματα όπλα που έχουν ε, τροποποιηθεί σε ήμι αυτόματα και θα μπορούσαν και ξανά να τροποποιηθούν σε αυτόματα. Επίσης θέλουμε να εξετάσουμε τα ημί αυτόματα για χρήση από τους ε, πολίτες ε, που έχουν μηχανισμούς αντίστοιχους ε, με τα αυτόματα, όπως είναι ένα ημιαυτόματο καλάζνικο, για παράδειγμα. Θέλω όμως να είμαι σαφής και πάλι. Υπό την υφιστάμενη οδηγία έχουμε ακόμα έξι κατηγορίες με αυτόματων όπλων, οι οποίες δεν τροποποιούνται από την πρότασή μας. Και είναι δυνατόν κάποιος ιδιώτης να τα αποκτήσει, βεβαίως ε, πάντα και σε συνάρτηση με τις εθνικές άδειες. Δεύτερη σημαντική πτυχή που θεωρώ σημαντική για την πρότασή μας για τα single weapons θεωρούμε ότι πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία, αλλά να καλύπτονται και από μια ενιαία άδεια. Και επίση προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τεχνικέ προδιαγραφέ για να διασφαλίσει ότι αυτά τα όπλα δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν σε πυροβόλα όπλα. Αυτό είναι το πρώτο σύνολο τροποποιήσεων σε ό,τι αφορά τι κατηγορίε πυροβόλων όπλων. Δεύτερο στοιχείο. Σε ό,τι αφορά τον παροπλισμό των ε, πυροβολών όπλων. Στο πλαίσιο της εφιστάμενης οδηγίας, τα παραπλεσμένα πυροβόλα όπλα δεν θεωρούνται πλέον πυροβόλα όπλα, αλλά απλά κομμάτια μέταλλο. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε ιδιώτης μπορεί να αποκτήσει αυτό το αυτό το, τα κομμάτια μετάλλου ε, οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οι πρόσφατες θερμοκρατικές επιθέσεις επιβεβαιώνουν ότι ορισμένα παραπλησμένα όπλα επανενεργοποιούνται και χρησιμοποιούνται από τους ε, τρομοκράτες. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Περιοπλισμό που υιοθετήθηκε στις 18 Νοεμβρίου εισάγει αυστηρότερα κριτήρια τα οποία θα περιορίσουν σημαντικά ε, τον, τον κίνδυνο της επανενεργοποίησης. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς αυτό τον κίνδυνο. Γι' αυτό στην πρόταση που υποβάλαμε προτείνουμε να απαγορεύσουμε την απόκτηση, την αγορά των πλέον επικίνδυνων πυροβόλων όπλων, ακόμα και μετά τον παροπλισμό τους. Αυτό αφορά την λεγόμενη κατηγορία Α. Ένα αυτόματο καλάσνικο, το οποίο έχει παροπλιστεί, για παράδειγμα, υπόκειται σε αυτή την κατηγορία, με βάση τη δική μας ε, πρόταση σε αυτό το στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις άλλες κατηγορίες πυροβολών όπλων, αυτές που δεν καλύπτονται από την κατηγορία Α, θα, μπορού, θα αυτά τα παραπλησμένα όπλα να τα αποκτήσει, να τα αγοράσει ένας ε, ιδιώτης, όμως προτείνουμε αυτά τα όπλα να υπάγονται στην απλή δήλωση. Το single declaration. Δεν θέλουμε ε, να δημιουργήσουμε επιπλέον φόρτο εργασία, διοικητικό άχθο, αλλά να, μπορεί να υπάρξει ε, σε περίπτωση ποινική ε, πράξη, αξιόπινη πράξη. Ε, μετά, η χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι κάτι το, ένα μέσο που χρησιμοποιείται ευρέω από τους ιδιώτε για την πώληση και αγορά όλων προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και των πυροβολών όπλων. Και γνωρίζουμε ότι η πώληση όπλων στο διαδίκτυο είναι κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελέγξει κανείς. Ξέρουμε όμως ε, ότι οι τρομοκράτες... Ε, αξιοποιούν αυτό το μέσο για να αγοράσουν ε, πλήρως παράνομα ε, ε, πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών. Οι συνάδελφοί μου, για παράδειγμα, τους πήρε πέντε λεπτά. Δεν τα αγόρασαν βεβαίως, αλλά βρήκαν στο διαδίκτυο ένα απλό πακέτο που επιτρέπει τη μεταφορά ενός ημιαυτόματου ή αυτόματου όπλου θεωρούμε ότι ο κίνδυνο για τους πολίτες είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επομένω, προτείνουμε να απαγορευτεί η αγορά ε, πυροβόλων όπλων από τους ιδιώτες στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ιδιώτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν όπλα από άλλο κράτος μέλος, όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσω αδειοδοτημένων, εξουσιοδοτημένων μάλλον ε, φορέων και εισαγωγέων. Τώρα για τους ε, εμπορευομένους και τους ε, συλλέκτε. Αυτή τη στιγμή αυτές οι κατηγορίες δεν υπάγονται στην υφιστάμενη νομοθεσία ε, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες διανομής τους. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω δυσκολίες για τους brokers και τους collectors, όμως θα πρέπει να υπάγονται στην οδηγία κατά τη γνώμη μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους απογορεύσουμε να αγοράζουν τέτοια όπλα, όμως θα πρέπει να ζητούν άδεια με τα ίδια κριτήρια, με τους ίδιους όρους όπως όλοι οι υπόλοιποι ιδιώτες. Τέλος. Αταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Οι πρόσφατε δημοκρατικέ επιθέσει έχουν καταδείξει τη σημασία τη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις που δίνονται σε ιδιώτες και τα κύρια χαρακτηριστικά των ε, όπλων. Αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο σε εθνικό επίπεδο. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα να μείνω εδώ για να σας δώσω δυνατότητα να παρουσιάσετε και εσείς τη σκέψη σχόλιά σας και ζητώ και πάλι συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ στην ώρα μου. Ευχαριστώ. Uh, Πρώτη σειρά ερωτήσεων από τους συντονιστές και μετά θα επανέλθουμε στα υπόλοιπα. Ερωτήσεις παρακαλώ και η Επιτροπή θα απαντήσει στη συνέχεια. Γκέπαρτ. ευχαριστώ, ευχαριστώ που μας ε, εξηγήσατε για μια φορά ακόμα τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί προφανώ ε, στην παρούσα φάση στο διαδικτύο γίνεται σωστή εκστρατεία. Άρα ως εκ τούτου καλό είναι να υπάρχει μια κάποια ηρεμία γιατί δεν στέκουν όλα αυτά που διαβάζουμε, που βλέπουμε και πολλά από αυτά που ζητούνται συνάδουν με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ακόμα νομοθεσία. Φυσικά θα πρέπει και το Κοινοβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο να τα εγκρίνουν. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προτάσεις που μας παρουσίασε μόλις η Επιτροπή, Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα χρειαζόμουν αρκετές διευκρινήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω το εξή. Το δεύτερο σημείο σε ό,τι αφορά τα όπλα συναγερμού θα πρέπει να αρκεί μια απλή δήλωση. Τι εννοείται όμως με τη δήλωση αυτή. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από την πρόταση αυτή που μας παρουσιάσατε. Για πείτε μας κάτι άλλο. Μία διευκρίνηση για τις ε, αγορές στο διαδίκτυο. Είπατε ότι δεν πρόκειται για παράνομο εμπόριο όπλων, αλλά στο τρίτο σημείο που αναφέρεται επανέρχεστε στο θέμα των παράνομων όπλων. Το κατανοώ ότι το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά είναι και θέμα ορισμού. Ποιος επιτρέπεται νόμιμα να αγοράζει τέτοια όπλα στο διαδικτύο. Δεν το κατάλαβα 100%. Γιατί από τις πρώτες προτάσεις που αναφέρατε, κατάλαβα ότι μόνο οι έμποροι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να αγοράζουν οι ιδιώτες, αλλά στη δεύτερη, τελευταία φράση, αν κατάλαβα σωστά, οι συλλέκτες θα μπορούν να αγοράζουν. Υπό ποιους όρους. Όμως, δεν θα θεωρούνται ιδιώτες, θα θεωρούνται εμπορευόμενοι. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Τελευταίο σημείο. Ανταλλαγή α, πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Αυτή η συζήτηση ήταν θυελώδης το 2008 όταν κάναμε την τελευταία τέτοια συζήτηση και τα κράτη-μέλη έδειξαν εξαιρετική απροθυμία να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύετε ότι δεδομένη τη ε, σημερινή κατάσταση ε, θα υπάρξει λίγο κάποια παραπάνω κατανόηση από πλευρά των κρατών μελών, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν απαραίτητο να ανταλλάσσονται πληροφορίε και διασυνοριακά για τον αριθμό, τον τύπο, την κατηγορία των όπλων, ποιο μπορεί να τα αγοράζει, να τα πουλάει. Γιατί οι κανόνε που έχουμε στα κράτη-μέλη διαφέρουν ασφαλώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κοινή νομοθεσία. Είναι σημαντικό λοιπόν το σημείο αυτό. Έχετε συζητήσει τα θέματα αυτά με τα κράτη-μέλη και θα είσαστε διτεθειμένοι να κάνετε το βήμα αυτό αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό. Okay. Um, just... Καλώς. οι συντονιστές ε, ε, δεν ξέρω, ε, ο Αντρές είναι εδώ, δεν ξέρω το ΕΛΚ ποιον θα προτείνει. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Απαιτείται αυστηρή νομοθεσία για τα όπλα αυτά. Έχουμε πανευρωπαϊκές αλυσίδες προσφοράς αυτών των προϊόντων Απαιτείται όμως οι νόμοι αυτοί να είναι λογικοί, να είναι εφαρμόσιμοι και να μην δημιουργήσουν μια παράνομη αγορά, γιατί την παράνομη αγορά δεν την ελέγχουμε. Και αυτά είναι τα όπλα που χρησιμοποιούνται στα εγκλήματα και στην τρομοκρατία. Δύο ερωτήσεις προς την Επιτροπή <clears throat> για τα εξουδετερωμένα όπλα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σε κυκλοφορία, δεν υπάρχουν αρχεία. Αν τα απαγορεύσετε από τη μία μέρα στην άλλη, θα αποσυρθούν και θα τα κρύψει ο κόσμος και δεν θα αλλάξει τίποτα. Ανησυχώ λοιπόν για τις προτάσεις. Τα εξουδετερωμένα όπλα εξορισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθεί και αν ενεργοποιηθούν εκ νέου τότε καθίστανται παράνομα. Αυτοί που έχουν ανάγκη από όπλα προφανώς θα αναζητήσουν άλλου είδους λύσεις. Έχετε αριθμούς για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί μέσω όπλων εξουδετερωμένων ε, και πραγματικά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ από τα μουσεία. Τι θα γίνει με τα όπλα που χρησιμοποιούνται στα μουσεία, <clears throat> τηλεόραση, κινηματογράφο, εκπαίδευση, κατάρτιση, ιστορικές αναπαραστάσεις. What is going to be the effect on them? Now, in terms of... Τι θα γίνει με όλα αυτά τα όπλα τώρα για τις πωλήσει τις διαδικτυακές. Πώς θα το ε, εφαρμόσετε αυτό. Συζητάμε το θέμα του διαδικτύου και της ενίας αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και ε, μήπως θα πρέπει να υπάρξουν νόμιμα σημεία πώληση έτσι ώστε ο κόσμος εφόσον έχει την άδεια να αγοράζει. Ε, δεν μπορεί κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο να αγοράσει online εκτός από την ελεγμένη άδεια κυκλοφορίας ε, όπλου ε, που θα δώσουν οι τοπικές αρχές. Λοιπόν, ας σκληρύνουμε την υπάρχουσα νομοθεσία για τους νόμιμους κατόχους, αλλά ας μην χειροτερεύσουμε την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε δύσκολες εμπειρίες με τα θέματα αυτά και νομίζω ότι οι νόμοι που ισχύουν είναι καλοί, είναι ε, σωστοί και δίκαιοι. Και οι προτάσεις της Επιτροπής θα υπονομεύσουν τα βήματα τα οποία έχουμε ήδη διανύσει. Σα ευχαριστώ, Πρέπει Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση τη. σύμφωνο ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα ναι, πιστεύω ότι το εμπόριο τέτοιων όπλων, ιδιαίτερα αποσυρμένων ε, όπλων είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει ασφαλώ όλα αυτά να ενταχθούν σε μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει στο διαδίκτυο και να αγοράσει ένα τέτοιο όπλο από οποιοδήποτε κράτο μέλο και να χρησιμοποιήσει τα εξαρτήματα για να φτιάξει ένα καινούριο όπλο. Και σε κάποιε περιπτώσει δεν χρειάζεται και καν ιδιαίτερη τεχνική γνώση για να γίνει αυτό. Σε ό,τι αφορά και τα απομεινάρια της ε, σύγκρουση στα Βαλκάνια, αυτό αποτελούσε ζήτημα και πριν από τις επιθέσεις στο Παρίσι, αλλά και τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι ήδη φυστάμενοι νόμοι εφαρμόζονται 100% και ότι δεν υπάρχουν νομικά κενά. Θα πρέπει να επιμείνουμε προκειμένου οι ελάχιστες προδιαγραφές, να τεθούν ελάχιστες προδιαγραφές για τα αποσυρμένα αυτό όπλα και κυρίως να εφαρμοστούν. Και γι' αυτό λοιπόν ορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόλα αυτά να προσέξουμε και να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η οδηγία και ποιος θα πρέπει να είναι πρώτος στο στόχος μας. Ε, θέλουμε να σταματήσουμε το παράνομο εμπόριο όπλων, αλλά να μην ε, τιμωρήσουμε παράλληλα και τους ε, πολίτες εκείνους που χρησιμοποιούν νόμιμα τα όπλα για ε, το κυνήγι για άλλους λόγους, για αυτό και να μην υπονομεύσουμε την νομοθεσία που υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη. Θα πρέπει οι πολίτες να μην θεωρήσουν ότι υπονομεύονται τα δικαιώματά τους. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στη διατύπωση που θα ακολουθήσουμε στην οδηγία, προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Άρα, το προτινόμενο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να καταστεί πιο συγκεκριμένο. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, και εγώ έχω λάβει εκατοντάδες email από τους ε, πολίτες της Τσεχίας και θέλω να εισακουστούν οι ανησυχίε τους και για την ε, συλλογική ασφάλεια, αλλά και για το σεβασμό των ε, ελευθεριών του πολίτη. Θα ήθελα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σαφής, ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη απαγόρευση μη αυτόματων όπλων. Το αναφέρατε αυτό. Για παράδειγμα, τα όπλα για αθλητισμό, για κυνήγι, θα επηρεαστούν από την πρότασή σας. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες θα ήθελαν να ξέρουν πιο πολλά για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε ασφαλώς ε, μετά τις εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη συζήτηση Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κάποιες φορέ έχω τη δυνατότητα ότι ακούμε τους πολίτες για κάποια ζητήματα, αλλά πολύ λιγότερο για άλλα θέματα, τα οποία όμως ε, είναι εξίσου σημαντικά και πολύ λυπάμαι γι' αυτό. Θα ήθελα να πω ότι η σύνδεση μεταξύ της ε, κατοχής ε, ε, και τη σχεδόν ελεύθερης ε, απόκτησης ε, όπλων με την ασφάλεια μας δείχνει ότι οι χώρες όπου είναι πιο ελεύθερη και πιο εύκολη απόκτηση τέτοιων όπλων είναι και η χώρα με 32.000 θύματα κάθε χρόνο εξαιτίας αυτών των πυροβολών όπλων. Στην Γαλλία είναι 365 θάνατοι κάθε χρόνο. Και δεν είμαστε και το παράδειγμα προς μίμηση, αλλά βλέπω ότι τα πάμε καλύτερα. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να θίξουμε ένα τέτοιο ζήτημα με τέτοια κλίμακα, ε, θέτοντα το μόνο στο πλαίσιο των ελευθεριών και ε, των συνηθισμένων κανόνων σε ό,τι αφορά το εμπορικό δίκαιο και την νομοθεσία. Κατανοώ ότι υπάρχουν οι κυνηγοί και μάλιστα κάποιος ε, έχασε τη ζωή του αυτό το Σαββατοκύριακο σε ένα δάσος επειδή πήγε για τρέξιμο και τον σκότωσε ένας κυνηγός κατά λάθος βεβαίως αλλά συνέβη. Υπάρχει και ε, ο αθλητισμός ε, στο πλαίσιο της... Η οπλοκατοχή στο πλαίσιο του αθλητισμού, όμως πρέπει να δούμε τι προεκτάσεις αυτό ενέχει για την νομοθεσία. Εγώ έχω υπηρετήσει και στο στρατό, επομένω είχα τη δυνατότητα να χειριστώ ζητήματα με αυτόματα μάλλον όπλα, όμω υπάρχει πολύ σημαντικό θέμα με την τροποποίηση των αυτόματων σε αυτόματα όπλα. Και αυτό βεβαίω ε, ε, φέρνει και έχει πολύ μεγάλου κινδύνους σε ό,τι αφορά και μαζικέ δολοφονίε. Είναι καλή δουλειά και σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί Προβλεπόταν βεβαίω γιατί έπρεπε να επανέλθουμε και στο κείμενο του 2008. Έχει κάνει η Κομισιόν τη, τη δουλειά που τη Όμω έχουμε και το ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είναι εξαιρετικά δραματικό. Θα ήθελα μόνο να μου πείτε, σε ό,τι αφορά τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κάποια κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δύο κατηγορίε όπλων. Τα, πυροβολ... τα απαγορευμένα όπλα και τα όπλα που υπάγονται σε αδειοδότηση. Ε, συνεχώς μιλούμε βεβαίως για το better regulation, να έχουμε μια νομοθεσία εύληπτη και κατανοητή από όλους. Ίσως εδώ λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να απλουστεύσουμε. Θεωρώ ότι αυτές οι 7-8 κατηγορίες όπλων είναι υπερβολικές. Γιατί λοιπόν να μην στραφεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ένα σύστημα με δύο μόνο κατηγορίες. Η μία κατηγορία που παίρνει άδεια και η άλλη που απαγορεύεται. Μετά άκουσα ότι πρέπει να ακούσουμε και τους ε, πολίτες που μας στέλνουν συνεχώς spam, mail ε, στους λογαριασμούς μας. Όμως ε, με ποιες ΜΚΟ ήρθε σε επαφή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, γιατί εγώ γνωρίζω το λόμπι των όπλων, θα ήθελα να μας πείτε αν και άλλα λόμπι ή άλλες οργανώσεις ήρθαν σε επαφή μαζί σας. Ήταν δύο ζητήματα που θέλω να θέσω απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. E Ο κύριο Ιβάσκοβιτς από το FDD. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Το προτινόμενο κείμενο, ιδίως ό,τι αφορά την ε, απαγόρευση των αυτόματων όπλων. αλλά και των ημιαυτόματων ή των ημιαυτόματων που μπορούν να τροποποιηθούν σε αυτόματα. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ημιαυτόματα όπλα και διερωτώ με κατά πόσο θα περάσουμε ακόμα και σε κατάσχεση όπλων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό μπορεί να επιφέρει και ζημίες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν γίνεται όλα αυτά να αιτιολογηθούν μόνο και μόνο με μια αναφορά στην ασφάλεια. Αυτό είναι μια διάσταση του προβλήματος έτερη διάσταση τώρα που με προβληματίζει. Η αιτιολόγηση της ε, αναθεώρησης της οδηγίας με την παραπομπή ε, αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων. Μήπως και αυτό είναι ένα λάθος ή και κάτι παραπάνω. Η νομοθεσία που θέλουμε να τροποποιήσουμε θα επηρεάσει ακόμα και τους νομοταγείς πολίτες, όχι τους τρομοκράτες. Ο νομοταγής πολίτης λοιπόν θα, δεν θα έχει εξίσου ευρεία πρόσβαση στα πυροβολά όπλα. Ανδρέας, θες να παρέμβεις. Πρόεδρε, πολύ λυπάμαι που έχασα την αρχή της ε, συζήτησης, αλλά χρειάστηκε να γυρίσω στο γραφείο μου λόγω τη καθυστέρηση τη άφεξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε νομίζω ότι ασφαλώς και το Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερο συμφέρον και ενδιαφέρον να υπάρχει μονονόμιμη κατοχή όπλων. Αυτό είναι λογικό και θα πρέπει κυρίω να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο η νομοθεσία που όντω να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ε, ε, έχουμε άλλα περιστατικά όπως τα πρόσφατα προσεκτικά. Νομίζω ότι και για τους κυνηγούς και για τους ε, όσους ε, για αθλητισμό χρησιμοποιούν όπλα δεν ε, περιλαμβάνονται τόσο πολύ στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο πολύ ενδεχομένως ε, προβληθήκαν στον τύπο. Αλλά γιατί, ε, αναρωτιέται ο τύπος, ε, γίνεται τώρα αυτή η τροποποίηση, αυτή η πρόταση δεν έχει να κάνει με τις τρομοκρατικές ε, επιθέσεις. Ήταν κάτι το οποίο προγραμματιζόταν εδώ και καιρό και Είναι σημαντικό νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει απόλυτα το ποιος είναι ο στόχος, ο σκοπός της ε, πρότασής της. Όσοι με νόμιμο τρόπο κατέχουν τα όπλα τους και τα χρησιμοποιούν για κυνήγι, για αθλητικούς σκοπούς, ε, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται. Εδώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια διευκρίνηση και νομίζω ότι αυτό θα κατεσυχασε και πολλές σχετικές ενώσεις κυνηγών και αθλητών στην Ευρώπη και μας προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα να σας διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών. Aloha Aho, Schwenfield, Dante, Karas, Metzola, and myself. So those, and Catherine Steiner, sorry. And you're, you're first. Um, um, so we have quite a lot of speakers. This... Έχουμε πολλούς ομιλητές και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσει το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και ζητώ συγγνώμη από τον προτέρων. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση αξίζει τον κόπο, γιατί ενδεχομένω να είναι και γρήγορε οι ερωτήσει αυτέ, σύντομε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντελσό για την παρουσίασή του. Στόχος της συζήτησης είναι το να κυνηγήσουμε τα παράνομα όπλα και να απαγορεύσουμε τα ημιαυτόματα που είναι πολύ ισχυρά και τα οποία μετασχηματίζονται εύκολα σε αυτόματα όπλα. Τώρα δεν θα τα συζητήσουμε τεχνικά αυτά. Η Επιτροπή κάνει μία πρόταση η οποία θα συζητηθεί στη Λίμπε και αφορά και τα παράνομα όπλα, το εμπόριο, το παράνομο εμπόριο των όπλων. Το Βέλγιο έχει πολύ σκληρούς νόμους, παρόλα αυτά πολλά όπλα πολλούνται παράνομα στις πίσω αίθουσες των καφενείων για ελάχιστα χρήματα. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Λοιπόν, έχει σημασία να δούμε ακριβώς τον εναρμονισμό ε, των ε, ρυθμίσεων ε, στις διάφορες χώρες. Πρέπει να υπάρχουν κοινέ διαδικασίες. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικά. Ε, θα πρέπει λοιπόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να εναρμονίσουμε με μία πρόταση οδηγίας. Γιατί όχι πρόταση κανονισμού. Με ένα συμβούλιο με 28 μέλη όταν θέλουμε να εναρμονίσουμε με οδηγία ε, καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν και όχι οφείλουν να. Συνεπώς λοιπόν κανονισμός. Και δεύτερον, και αυτό ακούστηκε ήδη, υπάρχει ένας τομέας που είναι η σκοποβολή, αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι επίσης, που θα πρέπει να είναι εκτός των ρυθμίσεων αυτών, εφόσον ε, εμπνευστούμε βέβαια από τις πιο προστατευτικές νομοθεσίες, μια εναρμόνιση προς τα άνω, και δεν θα πρέπει οι ε, αθλητές της σκοποβολής και οι κυνηγοί να είναι τα περιφερειακά θύματα μιας κατά τα άλλα θεμητής μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ Βίκη. Ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας, έδωσε, μας έκανε μια πρώτη παρουσίαση της πρότασης γιατί νομίζω ότι ε, πολλοί κόσμοι έχουν έρθει σε επαφή με τους ευρωβουλευτές και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και αρκετή σαφήνεια. Εκτιμώ τα όσα είπατε σε ό,τι αφορά την ρύθμιση για την απόκτηση και διανομή των όπλων, όμως δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε και τους πολίτες που νομίμως θέλουν να αποκτήσουν ε, όπλα, για παράδειγμα, για το κυνήγι. Τώρα, ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα δεν φοβάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, λόγω της έλλειψης επισημάνσεων για τα ημιαυτόματα όπλα οι αθλητικοί σύλλογοι, οι αθλητικές ενώσεις που αξιοποιούν τέτοια όπλα θα ζημιωθούν ε, χωρίς λόγο. Για παράδειγμα, κατανοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους προβληματισμούς ε, των νόμιμων ε, χρηστών όπλων. Μετά, στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται λόγος και για περιοδικούς ελέγχους με συμπληρωματική μαζικές επιστοποιήσεις στους κυνηγού, για παράδειγμα. Υπόθηκε ότι δεν μιλάμε για τα παράνομα όπλα, όμως ποια σύνδεση διαφαίνεται κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ των δύο για το γεγονός δηλαδή ότι οι τρομοκράτες ε, βρίσκουν παράνομα όπλα στα Δυτικά Βαλκάνια. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την εξαποστάσεως ε, αγορά όπλων στο διαδίκτυο για παράδειγμα, όταν έχουμε παράνομα όπλα στο διαδίκτυο, αυτό ήδη ε, θεωρείται πώληση από τις εθνικές αρχές ορισμένων κρατών μελών. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θεωρεί μια σοβαρή απειλή ε, σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους παράγοντες ελέγχου. Αυτό έχει νόημα, όμως το κείμενο αφορά κυρίως ε, τις πωλήσει μέσω διαδικτύου. Όμως, το ερώτημά μου αφορά τα, παράνομα, τα νόμιμα όπλα τα οποία διαφημίζονται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επομένω, με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει νόμιμη ε, πώληση, αγορά και πώληση αυτών των όπλων για, για τους κυνηγούς, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, I'm here and um, uh, uh, as Ευχαριστώ. Όπως ε, είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, όλοι κατανοούμε ότι Πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, πρέπει να υπάρχει νομοθεσία για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου όπλων. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι και το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό κάπου να τραβήξουμε τη γραμμή ούτω ώστε οι νόμιμοι κυνηγοί, όσοι ασχολούνται με τη σκοποβολή, και είναι και πολλοί αυτοί, δεν θα πρέπει να του απογορευτεί η δυνατότητα ε, να χρησιμοποιούν όπλα για τι νόμιμε αυτέ δραστηριότητε. Και πάλι λοιπόν, θα μπορούσατε να επαναλάβετε από πλευρά Κομισιόν ποια ή μη αυτόματα όπλα θα απαγορευθούν. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα, η αυτοματα οπλα θα απαγορευθουν αυτο ειναι το πρωτο δευτερον απο οτι καταλαβα η προταση σας αναφέρει κάθε πέντε χρόνια ε, να υπάρχει υποχρέωση ανανέωσης της άδειας και θα πρέπει να, για να δοθεί αυτή η άδεια να υπάρξει και σύμφωνη γνώμη ιατρού. Αυτό μου δίνει την εντύπωση ότι θα δημιουργήσει τεράστια γραφειοκρατία και οι γιατροί δεν θα έχουν το χρόνο να κάνουν άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Στη χώρα μου, τη Σουηδία, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην αστυνομία εάν κάποιος έρθει τους επισκεφθεί και για ιατρικούς σκοπούς δεν μπορεί να κατέχει όπλα. Στη Σουηδία αυτό δεν ισχύει μία φορά τα πέντε χρόνια. Οποιαδήποτε στιγμή κάποιο έρθει και κρίνει ο γιατρό ότι δεν θα έπρεπε να κατέχει όπλα, το αναφέρει στην αστυνομία. Είναι ένα καλό κανόνα για μα, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να προσθέσουμε και ένα επιπλέον επίπεδο γραφειοκρατίας. Αυτά προς το παρόν. Αλλά σας παρακαλώ να ακούσετε τις απόψεις μας και να μην προβούμε σε ενέργειες για την καταπολέμηση της δημοκρατίας που θα θίγει όμως τους δικούς μας νομοταγείς πολίτες. Εντάξει, εν συντομία έχουμε ακόμα νέο ομιλητές, δύο λεπτά έκαστος. Θα αξιοποιήσω το χρόνο που είχαμε για, την, ε, για το θέμα του ODR στις 6 το αργότερο. Επομένω, ε, θα είναι πιο σύντομη η συνεδρία των συντονιστών. Και αν δεν κλείσουμε αυτή τις 6.30 με τους συντονιστές θα δούμε τι θα κάνουμε με τη λίστα διάταξη της Πέμπτης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εντάξει. Κύριε Σαρλαλόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτής της πρότασης. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει πολλά σημαντικά στοιχεία για την ασφάλεια. Για παράδειγμα, ενισχυμένη συνεργασία. Πολύ θετικό αυτό. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων, η χνηλασιμότητα των όπλων και ούτω καθεξής. Και εγώ έλαβα πολλά mail σχετικά με αυτό το θέμα. Μέιλ που μου έχουν στείλει νόμιμοι κάτοχοι όπλων, ιδίως από την Τσεχία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική νομοθεσία. Ας εξετάσουμε τις περιπτώσεις χωρών που έχουν νομοθεσία υψηλής ποιότητας, όπου λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα. Υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει σχεδόν ε, καθόλου ε, πρόβλημα με τα παράνομα όπλα. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις ε, προσπάθειές μας στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου όπλων. Και εκεί να δώσουμε την έμφαση. Όμως, όπως είπε η Επιτροπή, το αντικείμενο της πρότασης δεν είναι τα παράνομα όπλα. Είναι καλές οι προσπάθειές μας, όμως δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε τους νόμιμους κατόχους όπλων. Γιατί από την νόμιμη οπλοκατοχή μπορούν κάποιοι να εξωθούν, να στραφούν μάλλον προς ε, τη μαύρη αγορά και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλους ε, κινδύνους και ως προς την ασφάλεια. Τώρα θέλω να κάνω τα εξής ερωτήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τα δικήματα που έχουν ε, διαπραχθεί με νόμιμα ή παράνομα όπλα. Έχει κάνει την αντιπαραβολή. Μετά σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, αυτή η παρανομα οπλα εχει κανει δυνατη παραβολη νομοθετική πράξη συνάδει και με την επιμέρους ε, εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και ποιο θα είναι ο συσχετισμό του, Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, ποια χώρα κατά τη γνώμη σα αποτελεί παράδειγμα προ μίμηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τα κατάφερε και ήρθε στις 18 Νοεμβρίου μας είχε παρουσιάσει ήδη κάποιες σκέψεις ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Σήμερα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μιλάμε για παράνομα όπλα. Τι μιλάμε, γιατί μιλάμε, γιατί συζητάμε. Μας αναφέρει παραδείγματα για παράνομο εμπόριο όπλων και τις σχετικές προτάσεις που θα κάνει. Όταν μιλάει για αποσυρμένα όπλα, τα οποία εκ νέου χρησιμοποιούνται παράνομα. Ασφαλώς αυτό δεν είναι νόμιμο όταν μιλάει για παράνομη απόκτηση όπλων στο διαδίκτυο αυτόματων όπλων ή μη αυτόματων όπλων. Μιλάμε για παράνομο εμπόριο και πραγματικά προκαλείται σύγχυση. Το είπε και ένας προηγούμενος ομιλητής. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε με τις καλές προθέσεις και να μην επανεφεύρουμε τον τροχό. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας για την καταχώρηση, την, ε, τον έλεγχο των όπλων. Δεν χρειαζόμαστε κάτι καινούργιο Έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, και φοβάμαι την, ε, τις επιπλέον γραφειοκρατικές ρυθμίσεις. Όταν Υπάρχει για παράδειγμα ένα σύστημα καταχώρηση όπως αυτό που έχουμε στην Αυστρία. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται ακριβώς. Και δυσκολεύομαι πως δεν θέλετε να πλήξετε του κυνηγού τους, ε, ε, ε, τις ενώσεις κτλ. Πώς θα το πετύχετε αυτό. Και αν ενημερωθείτε, θα ξέρετε ότι στην Ευρώπη μπορεί κανείς με 500 έως 1000 ευρώ να αγοράσει όπλα από σειράξεις παλιές. Μήπως, ε, λοιπόν, ε, καταλήγουμε στη διακριτική μεταχείριση των λάθος ομάδων των, του πληθυσμού. Δεν θέλετε, λοιπόν, να Υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση κάποιων ομάδων του πληθυσμού. Γιατί δεν ε, κάλεσατε λοιπόν στι διαβουλεύσει σα του κυνηγού, μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλα ε, μέλη τη κοινωνία για να ξέρετε τι κάνουν ακριβώ οι πρόεδρο. Ε. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και δυστυχά υπάρχουν κάποια στοιχεία στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δυστυχώ μα φαίνονται αμυγό ιδεολογικά και δεν συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της ιστορικής αγοράς ή σε μεγαλύτερη ασφάλεια και που θα επηρεάσουν αρνητικά πολύ μεγάλο αριθμό των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και τετέρως αναφέρομαι στην προτινόμενη απαγόρευση με αυτόματων όπλων. Πώς ε, μπορούμε να αποφασίσουμε κατά πόσο ένα ημιαυτόματο μοιάζει με αυτόματο ή δεν μοιάζει και σε τι βαθμό. Αυτά τα όπλα τα χρησιμοποιούν δεκάδε χιλιάδε σκοπευτές στην, ε, άτομα που ασχολούνται με τη σκοποβολή στην Ευρώπη. Έφεδρη. Σπανίως χρησιμοποιούνται για εγκλήματα και σχεδόν ποτέ για τρομοκρατικές ενέργειες. Τίποτα δεν υποδεικνύει ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφαλειά μας. Τα μη αυτόματα όπλα που μοιάζουν ε, με αυτόματα όπως το ΑΚ47 ε, είναι, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να μην μπορούν να μετατραπούν σε αυτόματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα με τα αυτόματα στα κριτικά όπλα ε, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις στο Παρίσι. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για κοινή όρη για την απόσυρση, για την ε, χρήση και την ε, διάδοση τέτοιων πληροφοριών. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα δικαιώματα των ε, πολιτών που ακολουθούν το γράμμα του νόμου δεν θα πρέπει να περιοριστούν χωρίς λόγο και ότι η απειλή της τρομοκρατία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για μια παράλογα και δυσανάλογη παραλογή και δυσανάλογη αντίδραση. Αυτό δεν θα προωθήσει το κύριο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πεπισμένος potrzebne. I niezależnie od tego, czy ότι ο κίνδυνος ε, υπάρχει. Ως εκ τούτου απαιτείται να υπάρξει ρύθμιση για την κυκλοφορία των όπλων, ανεξαρτήτως της χρήσεώς τους. Ο κανονισμός όμως αυτός θα πρέπει να είναι ε, λογικός και προσεκτικός, γιατί αλλιώς μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγικός. Οι ρυθμίσεις λοιπόν στις οποίες θα προχωρήσουμε δεν θα πρέπει να είναι αναποτελεσματικές και θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσει κανείς τα σύνορα ανάμεσα στην νόμιμη αγορά και στην παράνομη αγορά. Ε, στην νόμιμη αγορά ξέρουμε από πού πωλείται το όπλο μεν και πού αποθηκεύεται το όπλο, αλλά στις παράνομες συναλλαγές κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Εκεί όπου υπάρχουν απαγορεύσεις πάρα πολύ συχνά οι πολίτες ε, οι οποίοι θέλουν να σεβασμούν τον νόμο καταλήγουν σε φαιές ε, αγορές για να ικανοποιήσουν ε, τις ανάγκες τους. Διαρωτώ λοιπόν εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει σωστά ε, τις προτάσεις της και γνωρίζει πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα φυγούν από την συγκεκριμένη ρύθμιση. και επίσης τι είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες θα θυγούν και ποια είναι η αξία οικονομικά των προϊόντων για τα οποία μιλάμε. Η κυρία Στάινερ, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Μια και σήμερα συζητάμε τη χρήση των πυροβόλων όπλων ε, από τρομοκράτε και την απειλή στου Ευρωπαίου πολίτε Τα είδαμε αυτά στι φρικαλαιότητε του Παρισιού. Ξέρουμε εδώ και καιρό ότι υπάρχουν κάποια κενά στην νομοθεσία του 2008. Αυτά που προτείνονται λοιπόν εδώ προσπαθούν να καλύψουν ακριβώ τα κενά αυτά και την ανεχνευσιμότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών και γι' αυτό προτείνεται λοιπόν η συζήτηση αυτή να κοιτάξει ακριβώς πού έγκυται αυτή αυτά τα ελλείμματα, αυτά Σε ό,τι αφορά την πρόταση του 2008, 4,4 άρθρο, αναφέρεται ότι τα κρατημέλη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2000 Δεκεμβρίου θα εξασφαλίσουν την ε, ίδρυση και την εφαρμογή ενός ε, υπολογιστικού συστήματος, αποκριμένου συστήματος που θα δίνει πρόσβαση στα κράτη, στις αρχές σε ένα σύστημα για τα πυροβόλια όπλα και θα υπάρχει και διασυντική καταχώρηση. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει το άρθρο 4,4 και αναφέρονται και άλλα στοιχεία για την 20 ετία διατήρηση τέτοιων στοιχείων. Φυσικά, έχουμε και πιο αυστηρούς κανόνες, αλλά τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς θα πρέπει να εκτεθούν. Ένα δεύτερο ερώτημα για το κυνήγι. Κοιτάξα τις νέες προτάσεις και τις εφιστάμενες προτάσεις και δεν βλέπω να επηρεάζει κάτι το 12.2, το άρθρο 12.2. Αυτό μήπως απαντάει τις ανησυχίες των συναδέλφων. Πώς οι κυνηγοί χρησιμοποιούν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για τα όπλα που χρησιμοποιούν άσφαιρα. Ξέρουμε από τις συνομιλίες με τους αστυνομικούς αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καλύψουμε ως κενό γιατί δεν το κάλυψε η νομοθεσία του 2008. Ευχαριστώ. Και να σας ενθαρρύνω πραγματικά συνάδελφοι να πάτε στην αστυνομία να μιλήσετε με τους αστυνομικούς να δείτε τι συμβαίνει πραγματικά. Τώρα, στις διακοπές των Χριστουγέννων γιατί πιστεύω ότι θα μας ωφελούσε πάρα πολύ στη συζήτηση. Ντάντε. Ακούστηκαν πάρα πολλά και θα ήθελα δύο σημεία να υπογραμμίσω. Το πρώτο το οποίο θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να θέσουμε είναι η συζήτηση η οποία γίνεται για τη λεγόμενη νόμιμη αγορά δεν θα ήθελα να πιεστούμε έτσι ώστε να ερμηνεύσουμε την λεγόμενη νόμιμη αγορά με, με όρους σχετικούς και με θέματα όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εδώ το θέμα είναι η παράνομη αγορά. Η νόμιμη αγορά ελέγχεται ευτυχώς. Πρέπει να είμαστε εικονοποιημένοι. Έχουμε μια ελεγχόμενη αγορά με πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες ε, για την μη ευρεία κυκλοφορία όπλων που είναι πολύ επικίνδυνα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών. Ω εκ τούτου λοιπόν περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Επιτροπής ενδιαφέροντα στοιχεία όπως η ανιχνευσιμότητα, το θέμα της πιθανής απαγόρευσης της προμήθειας online τέτοιου είδους όπλων, όπως επίσης και ε, πυρομαχικών. Είναι βέβαια και κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν για να βελτιώσουμε την αγορά. Ε, αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε κάποια τέτοια όπλα να μην πέσουν στα χέρια των τρομοκρατών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προσπάθεια εναρμονισμού από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προς τα κράτη-μέλη τα οποία καλούνται να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο, εν περιπτώσει, ε, που να επηρεάζει ε, τις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Κατά τα άλλα, δεν πρέπει να διατρέξουμε τον κίνδυνο μιας ρύθμισης νομικής η οποία να θίξει τη ζωή πάρα πολλών συμπολιτών όπως των κυνηγών και των αθλητών στη, σκοτω... στη σκοπόβολη. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα, έχουν ένα ειδικό όπλο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα Ε, πραγματικά οι τρομοκράτες ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ορμούν με όπλα του 19ου αιώνα για να τελέσουν τις ε, πράξεις τους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την παράνομη κυκλοφορία των όπλων, το λαθρεμπόριο των όπλων. Αλλά θα πρέπει να μην δυσκολέψουμε τα όπλα που κινούνται στο εσωτερικό της νόμιμης αγοράς που ήδη ελέγχεται επαρκώς. Um, eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι μία σειρά σταθερών κανόνων με λογικούς στόχους και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος έλεγχος για την αγορά για τις αγοραπολισίες όπλων. Έχουμε να κάνουμε με ένα τμήμα της αγοράς το οποίο εντάσσεται στην ενιαία αγορά. Θα πρέπει όμως οι κανόνες οι αυστηροί που διέπουν τις συναλλαγές αυτές να ισχύουν και για τα πυρομαχικά, για τις σφαίρες. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρξει παρερμηνία των κανόνων. Οι πολίτες μας δεν θα πρέπει να νομίζουν ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί συνέβησαν αυτά τα οποία συνέβησαν στο Παρίσι. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε συνολικά τις τρομοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες Ξέρουμε τις ε, προσπάθειες που κάνουν οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες για να χρησιμοποιήσουν όπλα τα οποία να μην είναι ταυτοποιήσιμα, ανιχνεύσιμα και δεν θα πρέπει επίσης να θίξουμε τους αθλητές, τους κυνηγού, όπως επίσης και αυτούς που ασχολούνται με τα όπλα σε επίπεδο μουσιακό και συλλεκτικό. Έχω πάρει πάρα πολλά mail διαμαρτυρίας διότι υπάρχουν ανησυχίες για τον τρόπο εφαρμογής της συγκεκριμένης πρότασης και τον τρόπο επιρροής στους ανθρώπους, επηρεασμού μάλλον, των ανθρώπων που συλλέγουν όπλα ή που έχουν σαν χόμπι τα παλαιά όπλα. Θα συμφωνήσω λοιπόν με αυτούς οι οποίοι ε, θα ζητήσουν από την Επιτροπή να μάθουμε με ποιους ήρθαν σε επαφή εκ των προτέρων. Ότμα. Πρόεδρε, πολλά ακούσαμε και όλα υποδεικνύουν ότι υπάρχει μία ανασφάλεια. Ότι υπάρχει ανησυχία ότι πλήττονται οι λάθος άνθρωποι. Αυτό που είναι παράνομο είναι παράνομο. τα νόμιμα εύκολα μπορεί να θεωρηθούν παράνομα ή να γίνει κατάχρηση και να θεωρηθούν παράνομα. Υπάρχει ο κανονισμό, υπάρχει η οδηγία, υπάρχει και η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε. Η έκκλησή μου είναι να είναι πιο αντικειμενική η συζήτηση εδώ στην ε, Επιτροπή, γιατί οι πολίτες μας θα πρέπει να ξέρουν ότι τώρα ξεκινάει η συζήτηση στην Επιτροπή. Δεν είναι η τελευταία συζήτηση, πρόκειται για μια πρώτη ενημέρωση. Και μας έχει διευκρινίσει κάποια πράγματα αυτή η πρώτη ενημέρωση. Αλλά για να συνεχιστεί η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ξέρω κάποια πράγματα. Καταρχάς, θέλω να ξέρω τι γίνεται με την υφιστάμενη πρόταση για τις επιπτώσεις στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το εφιστάμενο δίκαιο στα κράτη-μέλη. Γιατί εδώ υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα και ποιότητε νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι επιπτώσεις για τι ε, αθλητέ, για τους κυνηγού, για τους συλλέκτε. Και τρίτον, θα ήθελα να ξέρω τι περιορισμοί θα σημαίνει αυτή η πρόταση για την νόμιμη κατοχή όπλων. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να ξέρουμε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης την γραμματεία της Επιτροπής τα email που έχουν λάβει τα μέλη της Επιτροπής να τα συνοψίσουμε και να τα υποβάλουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει απάντηση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, προς τα μέλη της Επιτροπής και να μην χρειαστεί να απαντάει ο καθένας μας ξεχωριστά, να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υπάρχει και ένας μπούσουλας για την κοινοβουλευτική μας εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλάς. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα έθεσαν οι συνάδελφοι. Έχω ένα άλλο ερώτημα όμω. Πάντα λέμε εδώ ότι η νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε μελέτες και αναλύσεις. Και έτσι έχουμε αυτή την έκθεση που βασίζεται ε, σε μία μελέτη αξιολόγησης. Όμως δεν έχουμε λάβει, λάβει υπόψη ορισμένα στοιχεία, μόνο την κατηγοροποίηση των όπλων. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ της μελέτης ε, και της ε, πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, ζητώ από την Κομισιόν να διευκρινίσει σε τι είδου συστάσει βασίζεται η πρότασή τη. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μία μικρή παρατήρηση. Το 2008 οι συνάδελφοί μου εξέτασαν την αναθεώρηση τη οδηγία. και η τελική διατύπωση ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει με τις διαδικασίες το 2013 κτλ. Θα εκδώσει κατητήριες γραμμέ ε, για τι ε, δυνατότητε και διαδικασίε απόσυρσης, ούτω ώστε αυτά τα όπλα, τα αποσυρθέντα, τα εξωτερωμένα, να μην μπορούν πλέον να επανασυμποποιηθούν. Αυτό το 2008. Εφτά χρόνια μετά, το 2015, επιτέλους δημοσιεύσατε αυτές τις κατητήριες γραμμές. Οι συνάδελφοί μου, υποθέτω, ότι θα θέλουν να υπάρξει απείρως περισσότερη σαφήνεια για το τι θα συμβεί στο μέλλον, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα ζητήσουμε θα γίνει πραγματικά και θα υπάρξει πραγματικά ξεκάθαρη και σαφής διατύπωση. Είχατε πει αρχικά ότι δεν θέλατε να απαγορεύσετε όλα τα μη αυτόματα όπλα, γιατί όσα ήταν στην κατηγορία Β θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα. Όμως αυτό δεν είναι για μένα σαφές Διαβάζοντα κανεί την πρόταση και μάλιστα στη μετρική μου είναι γραμμένη αυτή η πρόταση. Φανταστείτε τι θα καταλάβουν οι υπόλοιποι προσπαθούν να τη διαβάσουν. Το resemble που λέτε εσείς στην πρότασή σας, το προσωμιάζουν, είναι ιδιαίτερα υποκειμενικός όρος. Επομένω, θα μπορούσατε να διασκεδάσετε ορισμένες ανησυχίες, εάν δείτε με μεγάλη προσοχή ποιες είναι οι προθέσεις σας και προσπαθήστε στη συνέχεια να καταλήξετε σε μια καλύτερη διατύπωση, καλύτερη χρήση της αγγλικής, ούτως ώστε πραγματικά αυτά τα όπλα να μην μπορούν πλέον να επαναχρησιμοποιηθούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο ε, εν συντομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσει στο μέλλον. Θα μιλήσουμε με του συντονιστέ, πότε θα διοργανώσουμε ενδεχομένω και ξεχωριστέ συζητήσει. Μάλιστα. Θα είμαι σύντομο γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει και πολλή χρόνο. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα νόμιμα όπλα, 10.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους ε, την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη με τη χρήση νομίμων όπλων. Είναι πραγματικό πρόβλημα λοιπόν. Αν δείτε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, δεν χρησιμοποιούσαν παράνομα όπλα, όπλα ε, νόμιμα όπλα συγγνώμη, χρησιμοποίησαν. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα λοιπόν. Δεν είναι τεχνητό. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, κάνουμε αυτή την πρόταση βάσει ξεχωριστών συζητήσεων, μελετών και αναλύσεων με όλα τα διαφέρμενα μέλη. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς ε, επινοήσαμε. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας. Πράγματι, και η χρονική συγκυρία επιτάχυνε τις διαδικασίες. Τα γνωρίζετε. Τρίτο στοιχείο, για τους κυνηγού. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Το κείμενο παραμένει ως έχει. Αν δείτε το παράρτημα 1 βλέπετε ότι η κατηγορία Γ δεν επηρεάζεται στο παραμικρό από αυτή την πρόταση. Δεν αλλάζει τίποτα λοιπόν. Για την κατηγορία Β που αφορά κυρίως, ε, μάλλον τους κυνηγού, αλλά κυρίως ε, όσους ασχολούνται με την αθλητική σκοποβολή. Στην κατηγορία Β λοιπόν, που υπάγεται στην αδειοδότηση, μπορεί κανείς α μάλλον τέσσερα. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ή μη αυτόματα όπλα με θαλάμους ε, και πυρομαχικά για τρεις γύρους συνολικά. 40 κάτι σφαίρες. Όλα αυτά δεν επηρεάζονται από την πυρότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένω, όσοι ασχολούνται με την αθλητική σκοποβολή δεν θα επηρεαστούν, θα εξακολουθήσουν να ασχολούνται με το χόμπι τους. Αυτό που απαγορεύουμε είναι τα ημιαυτόματα όπλα που μοιάζουν με αυτόματα. Πράγματι το resemble μπορεί να μην είναι αρκετά σαφής Τα γλυκά σας βεβαίως και είναι καλύτερα τα δικά μου. Ε, αλλά είναι και μια διαδικασία διαβουλεύσεων ε, με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο. Μπορούμε να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση. Όμω, για να είμαστε σαφεί, κατά νου έχουμε τα καλά καλάζνικοφ, για παράδειγμα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δολοφονίε, για παράδειγμα. Και αν μου λέτε ότι οι κυνηγοί και οι ε, αθλητικοί σκοπευτέ χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα, τότε μπορεί να υπάρχει διαφωνία μεταξύ μας να το συζητήσουμε. Όμω βλέπουμε ότι στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο εύκολο να βρει κάποιο ένα ημιαυτόματο που μπορεί να το κάνει αυτόματο. Αυτό υπάρχει και είναι πολύ συνήθες. Αυτό θα επηρεαστεί. Όμω θέλουμε και θα δεχτούμε οι κυνηγοί και οι σκοπευτέ να αξιοποιούν αυτά τα όπλα. Αυτό είναι δική σα επιλογή. Για τη διατύπωση και τα λοιπά, εντάξει πράγματι μπορούμε να τα βελτιώσουμε ενδεχομένω. Εν συντομία να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια, δεν θα απαντήσω σε όλα, δεν είναι δυνατόν. Πράγματι, χρειάζεται να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Είναι πλέον διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να ε, προβούν σε αυτήν την ανταλλαγή δεδομένων. Και κάτι τελευταίο ε, για την απόσυρση εξοδετέρωση των όπλων. Θέλουμε να διευκρινίσουμε την κατάσταση και το έχουμε κάνει σε έναν βαθμό με τα εκτελεστικά μέτρα που υιοθετήσαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Θα μείνω εδώ γιατί ξέρω ότι πολλά σημεία ακόμα εκκρεμούν. Ευχαριστώ πολύ. Η Γραμματεία θα ήθελα να κατατήσει μία σύνοψη όλων των ζητημάτων ε, που αναφέρθηκαν και να σας θυμίσω ένα από τα κύρια ζητήματα ε, που θίξατε. Θα συζητήσουμε και με τους συντονιστές τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για ε, να εισακουστούν όλες οι απόψεις και επιθυμίες όπω συμβαίνει και με όλου του νομοθετικού φακέλου, τα μέλη μα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσει ε, για την τροποποίηση τη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. To give us a presentation on the state of play of the... Παρουσίαση ε, για την ε, επιγραμμική επίλυση διαφορών. Η κυρία Δεσμίνα Σπανού. Would you like to start? Θα ξεκινήσεις. Thank you. Um, hello, Madam Chair. I Να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε. Εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε σε αυτή την Επιτροπή να σας πούμε τι συμβαίνει με την πλατφόρμα των επιγραμμικών επιλύσεων διαφορών. Ε, φτάνει η ώρα της ε, έναρξης, όπως ξέρετε, και ο κανονισμός ε, πρέπει να είναι έτοιμο ε, μέχρι τι 9 Ιανουαρίου του 2016. Ήδη έχει γίνει μια παρουσίαση για τα μέλη της Επιτροπής. Σήμερα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το πώ έχει η κατάσταση σήμερα και να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία στοιχεία. Ε, κατανοώ ότι δεν υπάρχει πολλή χρόνος. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία ε, που δημοσιεύθηκαν το Σεπτέμβριο σχετικά με την άποψη καταναλωτών και εμπορευομένων σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό εναλλακτική επίλυση διαφορών και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Βλέπετε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό το μέσο. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτέ στι διασυνοριακέ του αγορέ, μία στι τρει, είναι ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν ξέρουν πώ να επιλύσουν και αν θα είναι σε θέση να τα επιλύσουν. Ιδίω αν ο εμπορευόμενο είναι σε άλλο κράτο ε, δεν κινούν άλλε διαδικασίε γιατί είναι μικρό το ποσό ή φοβούνται ότι θα είναι μακρά η διαδικασία επίλυση. Θεωρούμε ότι το ODR μπορεί εδώ πραγματικά να κάνει διαφορά. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι 45% των καταναλωτών θεωρούν ότι είναι εύκολο να λύσει κάποιο ε, τι διαφορέ μέσω του ADR και 70% δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη χρήση του ADR. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το γνωρίζουν οι εμπορευόμενοι είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά άγνοιας ή απροθυμίας. Το 50% θεωρεί ότι δεν είναι διαθέσιμο στον κλάδο του, γι' αυτό και δεν καταφεύγει σε αυτόν τον μηχανισμό. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο, το έχουμε προσθέσει και στο παρελθόν, έχουμε ένα πακέτο, ε, την οδηγία τη εναλλακτική επίλυση διαφορών που υποτίθεται ότι τα κράτη-μέλη θα, θα είχαν μεταφέρει μέχρι τα, τον Ιούλιο τρέχοντος. Ότι θα υπάρχουν δηλαδή αντίστοιχε οντότητε, αντίστοιχοι φορεί ε, για όλου του κλάδου. Και το δεύτερο τμήμα του πακέτου, κανονισμό για την επιγραμμική πλατφόρμα επίλυση διαφορών, που αφορά όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις γλώσσες, το οποίο έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί με την, υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσφέρει συνδρομή σε όλα τα κράτη-μέλη τι θα μας φέρει αυτό το πακέτο. Μία νέα νοοτροπία εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών, πιο απλή, γρήγορη και ε, λιγότερο δαπανηρή διαδικασία. Θα υπάρχει ένα ποιοτικό σύστημα, θα υπάρχει δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, αλλά ε, θα αυξηθεί και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό θα θέλαμε να σα παρουσιάσουμε σήμερα. Τώρα, στη αφορά την ε, μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Μέχρι τώρα 14 κράτη-μέλη έχουν ολοκληρώσει τη δικασία μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τη οδηγία. Ε, κάποια κράτη-μέλη, 8 τον αριθμό, έχουν μεταφέρει μερικώ ε, την οδηγία και θέλουν να έχουν ολοκληρώσει τη δικασία μέχρι τον Ιανουάριο. Όμω δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα, θέλω να σα πω, γιατί συνήθω υπάρχουν μεγαλύτερε καθυστερήσει. Επομένω, ε, νομίζουμε ότι έχουν πάει καλά τα πράγματα. Πολλά έχουν μεταφέρει την νομοθεσία και έχουν κοινοποιήσει και τους ε, φορείς ADR. Ε, κάποια κράτη-μέλη δεν θα ολοκληρώσουν η δικασία μέχρι, τους επόμενους, μέχρι τη λήξη προθεσμίας στους επόμενους μήνες, είτε λόγω κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Ένα μικρό αριθμό λοιπόν δεν θα τα έχει καταφέρει, αλλά ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι του 2016 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για την ε, κοινοποίηση των ε, φορέων ADR. Η, νομοθεσία, η προθεσμία θα ήταν ε, η ίδια με την θέση σε ισχύ τη πλατφόρμα. Ήταν ένα πρακτικό πρόβλημα το οποίο είχαμε προβλέψει, ζητώντα τα κράτη-μέλη να κοινοποιήσουν πριν από την προθεσμία. Η Επίτροπό μα, κυρία Γιούροβα, έχει ε, αποστείλει επιστολέ σε όλα τα κρατημέλη και έχει πείσει αρκετά κρατημέλη. Οι περισσότεροι λοιπόν θα στείλουν τον κατάλογο πριν από την προθεσμία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα ODR, πώς έχει η κατάσταση. Ξέρετε ότι κινούμαστε εντό χρονοδιαγράμματο. Έχουμε προετοιμάσει όλο το τεχνικό σκέλο, γιατί ξέρουμε ότι τον Γενάρη είναι η προθεσμία. Όμω δεν μπορεί να λειτουργήσει μια πλατφόρμα εάν δεν συνδέεται με τι ε, σχετικέ ε, αρχέ ADR και πάλι θεωρούμε ότι στις αρχές του 2016 θα υπάρχει επαρκή σκάλυψη. Σε ό,τι αφορά τους εμπορευόμενους, να υπενθυμίσω ότι υποχρεούνται από την νομοθεσία να έχουν link που να παραπέμπει στο ODR στον ιστότοπό τους. Τι περιμένουμε λοιπόν η προθεσμία ήταν η 9η Ιανουαρίου, αλλά όπως ε, προανέφερα δεν αναμένουμε ότι θα είναι έτοιμα τα μέλη. Γι' αυτό σκεφτόμαστε να μεταφέρουμε ε, την έναρξη στις 15 Φεβρουαρίου, γιατί μέχρι τότε θεωρούμε ότι θα υπάρχει μια κρίσιμη μάζα 100 μελών που θα έχει συνδεθεί με το σύστημα, περίπου 20 ίσως και παραπάνω γιατί είναι σημαντικό όταν πάει ο πολίτης στον ιστότοπο να λύσει το πρόβλημά του, να μην απογοητεύεται γιατί βλέπει ότι το κράτος μέλο του δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Η επίτροπο προτείνει λοιπόν να μεταφερθεί η ένταξη για τις 15 Φεβρουαρίου, που και πάλι βρίσκεται στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας και ε, τότε θα τεθεί ε, στη διάθεση του κοινού η πλατφόρμα. Θέλουμε από τις 9 Ιανουαρίου να ξεκινήσουν δοκιμαστικές ε, λειτουργίες, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Βεβαίως, ε, βασιζόμαστε και σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού να προβάλλουν το EDR από τι αρχέ τη χρονιάς. Είναι σημαντικό να ενημερωθεί ο πολίτης ε, για αυτή την εξέλιξη. Επομένω, πρέπει να υπάρξει και η δική σα συνεργασία για την επιτυχή έναρξη του προγράμματος στι 15 Φεβρουαρίου. Τώρα, πώ λειτουργεί η πλατφόρμα. Ήδη το ελέγξαμε και το παρουσιάσαμε στην ΙΜΚΟ. Είναι όμω η πιο πρόσφατη παρουσίαση τη πλατφόρμας αφορά τους τέσσερις χρήστες, ο καταναλωτής που κάνει την ένσταση, ο εμπορευόμενος που ανταποκρίνεται, η αρχή που χειρίζεται την κατάσταση και τέλος το σημείο επαφής ε, που συνδράμει όλους τους χρήστες καθόλου τη διάρκεια της διαδικασίας. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Και η διαδικασία έχει τέσσερα σημεία, υποβολή ε, του παραπώνου, ε, συμφωνία με την οντότητα EDR, διαχείριση της υπόθεσης από την αρχή EDR και το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης. Βλέπετε ότι πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό, διαφορετικό, καινοτόμο. Πρώτα, ο καταναλωτής δίνει τα στοιχεία του εμπορευομένου. Α, προχώρησα πολύ. Αυτή τη μορφή έχει, μάλλον αυτό είναι το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσει ο καταναλωτής κάποια στοιχεία θα συμπληρώνονται για αυτομάτω. Μετά ο καταναλωτή πρέπει να περιγράψει την υπόθεση, τι αγόρασε, με ποιο αντίτιμο, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετώπισε και μετά να δώσει τα στοιχεία του. Όταν συμπληρωθούν αυτά τα στοιχεία, ο καταναλωτή υποβάλλει το παραπονό του, το οποίο μεταφέρεται στον εμπορευόμενο. Είναι λοιπόν πολύ γρήγορη και αποτελεσματική η διαδικασία. Αυτό λαμβάνει ο εμπορευόμενο. λοιπόν μία κοινοποίηση ότι έχει γίνει για εσάς ε, ένα παράπονο, μια καταγγελία ε, και θα αποφασίσει αν θα συμφωνήσει να προχωρήσει με αυτή την ε, εξοδικαστική διαδικασία. Τότε θα πρέπει να δώσει τη δική του εκδοχή της υπόθεσης ε, και να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε φορέα ADR που είναι συνδεμένο με το σύστημα. Σε ευρωπαϊκή βάση είναι σημαντικό. Όταν συμφωνήσουν και οι δύο επί της αρχής ADR, η υπόθεση μεταφέρεται, διαβιβάζεται απευθεία σε αυτή την αρχή. Εδώ βλέπετε... Α, συγγνώμη, από μόνο του προχωράει με τις διαφάνειες. εδώ βλέπετε μία απεικόνιση της ε, αρχής της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που λαμβάνει την υπόθεση και με τις δύο εκδοχές, του καταναλωτή και του εμπορευομένου έχει διάφορε λειτουργίε για να διευκολύνει τη διαχείριση τη υπόθεση, ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των δύο μερών, ε, διαχείριση και έκδοση τελική απόφαση που διαβιβάζεται στα δύο μέρη. Και εδώ βλέπετε την τελική εικόνα για όλες τις υποθέσεις και διασωνηρακά αυτή την εικόνα θα έχει πάνω κάτω η πλατφόρμα. Θέλαμε να σα τη δείξουμε. Την έχουμε δοκιμάσει δύο φορέ με όλα τα διαφορετικά μέρη και εδώ στι Βρυξέλλε, αλλά και άλλη φορά σε διαφορετικέ χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαφορετικά σενάρια, άνθρωποι που την μπήκαν δηλαδή είτε ω καταναλωτέ είτε ω εμπορευόμενοι, είτε ω αρχέ και ήταν πολύ επιτυχής αυτέ οι δοκιμέ. Λάβαμε υπόψη όλα τα σχόλια και αυτή είναι η τελική μορφή τη πλατφόρμας. Έχουμε λάβει και πολύ θετικά σχόλια γιατί θεωρείται εύχριστη πλατφόρμα και ελπίζουμε ότι και εσείς την ίδια γνώμη θα έχετε. Και είμαστε διατεθειμένοι να την παρουσιάσουμε και πάλι όποτε το επιθυμείτε. Θα έχουμε δοκιμές όλο τον Ιανουάριο πριν ξεκινήσουμε επισήμως στις 15 Φεβρουαρίου. Σας έκανα αυτή την πολύ σύντομη παρουσίαση γιατί μου είπατε ότι δεν υπάρχει και πολλής χρόνος με τα χαράς να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Very ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, πολύ συνεκτική αυτή παρουσίαση και νομίζω εκτιμούμε ιδιαίτερα την δουλειά που κάνατε για να πραγματοποιηθεί αυτή η παρουσίαση. Οι συνάδελφοι, ποιοι θέλετε να θέσετε ερωτήσεις. Δεν βλέπω κανένα να θέλει να κάνει ερώτηση. Εγώ έχω μια ερώτηση να κάνω εφόσον μου επιτρέπετε. Έχουμε 14 που έχουν εφαρμόσει μερικώς ε, την, ε, το, το μηχανισμό αυτό. Ποια ήταν τα βασικά εμπόδια. Υπήρχαν ζητήματα συγκεκριμένα, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν κάποια συστήματα ειδικά και να έχουν εφαρμοστεί, γιατί νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μεγάλο όγκο εργασία εδώ και εμεί εκπροσωπούμε και τα 28 κράτη-μέλη. Αν θέλετε να απαντήσετε, ναι, πολύ καλό ερώτημα. Καταρχάς, ο θεματοφύλακας της, ε, των συνθήκων, αυτό που κάναμε ήταν να αποστείλουμε επιστολές μετά την παρέλευση της ε, καταληκτικής ημερομηνίας στα κράτη-μέλη που δεν είχαν εφαρμόσει την νομοθεσία. Απάντησαν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό καταδεικνύει πόσο σοβαρά παίρνουν ε, τα κράτη-μέλη αυτό το έργο. Ένα τέτοιο θέμα λοιπόν ήταν και η πλατφόρμα ODR και τα προβλήματα που υπάρχουν για τα κράτη-μέλη όπου το σύστημα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να δημιουργηθούν και τα σχετικά κριτήρια που προαπαιτεί η νομοθεσία προκειμένου να δημιουργηθούν αυτές οι οντότητες ODR ε, ή να αναβαθμιστούν. Αυτό ασφαλώς παίρνει χρόνο. Έχουμε τρία-τέσσερα κράτη-μέλη όπου υπήρχαν εκλογές και υπήρχαν νομοθετικά ζητήματα τα οποία ανέκυψαν και δεν ε, τους επέτρεψαν να ολοκληρώσουν την εργασία μέσα στην προθεσμία. Υπήρχαν λοιπόν αντικειμενικοί λόγοι, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ε, ευκαιρία να έχουμε συγκεντρώσει μια κρίσιμη μάζα μέχρι το Φεβρουάριο και όλοι νομίζω θα το έχουν εφαρμόσει μέχρι το καλοκαίρι. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος για τη διευκρίνηση αυτή. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από πλευρά των συναδέλφων, ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση που ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική και έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη. Και τώρα ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών.